Chers collègues, je vous suggère de... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις εργασίες μας γιατί έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Και έχουμε μια γνωμοδότηση την οποία δεν κάναμε χτες ε, στην στιγμή που έπρεπε. Περνάμε στο ψήφισμα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους. Αυτό μετά από την ε, δολοφονία του συναδέλφου Νταμί. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο για την, ε, το ψήφισμα αυτό. Ε, Ο κύριος Πίτερ Κάιζερ πρώτα απ' όλα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω το ότι η Επιτροπή των Περιφερειών αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία η οποία είναι αναγκαία και δείχνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο το μίσος και τη ρητορική μίσους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και βλέπουμε συνεχώς τέτοιες περιπτώσεις αλλά και δολοφονικές απόπειρες. Γι' αυτό Θεωρώ ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν μια κοινή πρωτοβουλία κατά του μίσου στο διαδίκτυο. Οι νομικές συνέπειες είναι το ένα, αλλά χρειαζόμαστε και προληπτικά μέτρα στον τομέα της ε, ευθύνης ε, των ΜΜΕ, του σχηματισμού συνειδήσεως ε, στα σχολεία και στις ενώσεις. Δεν επιτρέπεται να έχουμε μια κοινωνία η οποία επικοινωνεί μόνο μέσω του μίσου στα κοινωνικά μέσα. Χαιρετίζω το ότι η Επιτροπή των ε, Περιφερειών απευθύνει έκκληση σε όλους τους υπεύθυνους αφενός την ίδια την πολιτική να καταργηθεί να, και να καταδικάσει το μίσος και τη ρητορική μίσους αλλά Απευθύνω επίσης έκκληση. Εκεί όπου μπορούν να ληφθούν μέτρα θα μίμιε στην δικαιοσύνη να υπάρχει συνεργασία, κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα που ξεκινήσαμε στην Αυστρία στην Ένωση των Δημάρχων όπου προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε το μίσος στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ λοιπόν ρητός για το ότι η Επιτροπή των Περιφερειών αναγνωρίζει πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το μίσος με όλες τις νομικές δυνατότητες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριος, κύριος Βόσνιγκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επωφεληθώ της ευκαιρίες που μου δίδεται και να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να εγκριθεί αυτή η πρόταση για να φτάσουμε στο σχέδιο ψηφίσματος σήμερα. Πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι ότι το πολύ σημαντικό για να θυμηθούμε τον συνάδελφο Πάβελ Ανταμόβιτς και κυρίως για να μπορέσουμε να κάνουμε ως Επιτροπή των Περιφερειών δημόσια αυτή την συζήτηση τόσο σημαντική. Γι' αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι η καταπολέμηση ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους. Θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα ένα στοιχείο που κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα θα πρέπει να τα μελετάμε εκ των υστέρων και να συλλογιζόμαστε πραγματικά σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε μετά από τέτοιου είδους πράξεις. Και εδώ συμπεριλαμβάνονται τέτοιου είδους συμπεράσματα. Για μένα είναι σημαντικό να δούμε ποιος πρέπει να επομιστεί την ευθύνη για τέτοιου είδου γεγονότα. Οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε πρότυπα. Όταν κάποιος ενεργεί με μίσος στρέφει τη συμπεριφορά του και την πράξη του κατά ενός πολιτικού, όπως τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά επιτίθεται συγχρόνως και κατά της πολιτικής, κατά όλων των πολιτικών. Είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας και ελπίζω ότι θα μπορέσει να αποτελέξει βάση σκέψης και άξονα που θα κατευθύνει τον τρόπο που θα σκεφτόμαστε για όλους και θα είναι μια πολύ καλή υπενθύμηση του τι ακριβώς συνέβη στο συνάδελφο. Αυτό προς το καλό όλων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάτεν έχει το λόγο. Κυρία Γιάτεν, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος Ολλανδικής Αντιπροσωπείας θα ήθελα να πω πως το ψήφισμα αυτό οφείλεται σε κάποια θλιβερά γεγονότα. Βεβαίω τα είχαμε και στην Ολλανδία. Ε, είχαμε δολοφονίε πολιτικών. Ο ένα ήταν ο Πιμ Φορτάιν και ο άλλο ο κύριο Φανχόχ και άφησαν βαθιέ πληγέ στην χώρα. Ακριβώ λοιπόν. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι απέναντι σε αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά ανώνυμα στο διαδίκτυο. Και πρέπει να στείλουν το σωστό μήνυμα εδώ, Δήμοι και Περιφέρειες όλοι οι πολίτες ενωμένοι. Αλλά θα πρέπει οι πολιτικοί να μπορούν να διοικούν ασφαλείς ε, χωρίς ε, να φοβούνται για την ζωή τους στην Ολλανδία. Οι απειλούμενοι δήμαρχοι κέρδισαν το βραβείο Μακιαβέλη. Βεβαίω είναι ένα βραβείο το οποίο δεν θέλει κανεί να κερδίσει, γιατί είναι ένα βραβείο που κερδίζουν όταν τον απειλούν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε ε, για το ψήφισμα αυτό. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι και να δημιουργήσει κάποια α, συνείδηση ε, για το ότι όσοι κάνουν τέτοια πράγματα ανωνύμως και ήμι ανωνύμως μπορούν να έχουν και να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες. Σας ευχαριστώ κύριε Μπριγκίτ Χονέ. Ε, ευχαριστώ και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό αυτό το ψήφισμα. Βλέπουμε τους κινδύνους της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους και θα πρέπει ακριβώς οι πολιτικοί να καταπολεμήσουν την ε, ε, πολιτική αυτή στην ε, κοινωνία και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες ε, που είναι ενεργητικά υπέρ της ανεκτικότητας και κατά του μισού και αυτό πρέπει να αναφερθεί στο ψήφισμα γιατί πρέπει να είμαστε μαζί τους στην πρώτη γραμμή. έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία και θα ήθελα να τη στηρίξετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ορτήλ έχει τον λόγο. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ε, Szanowni państwo, popieramy tę rezolucję, uważamy ją za ważną. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Πιστεύουμε ότι είναι και πολύ καλό και απαραίτητο στην παρούσα στιγμή. Πρόκειται για ένα ψήφισμα που μας κάνει να θυμηθούμε τους αντικειμενικούς στόχους της Ευρώπης. Στόχους στους οποίους μπορεί να πλήξει κάποιος με τη συμπεριφορά του. Επίσης, θα θέλαμε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον συνάδελφο Αντάμοβιτς να περάσουμε το ψήφισμα αυτό και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας τα ένθερμα σε όλους τους οικείους τους. Οι δολοφόνοι ξέρουμε ότι είναι άρρωστοι. Δεν πρέπει κανείς ε, να περιορίζεται λέγοντας ότι πρόκειται για πολιτική πράξη. Πρέπει να βασιζόμαστε στα γεγονότα, στην ε, αλήθεια και να μην αφήνουμε την παρεκτροπή κάποιων οι οποίοι οδηγεί σε τέτοιου είδους απεχθείς πράξεις. Θα πρέπει ως κοινωνίες να αναλύουμε τα γεγονότα, να αρχίσουμε να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τα μέσα ενημέρωσης, με ποιο τρόπο μεταφέρουν κάποιες ειδήσει. Τα μέσα ενημέρωση τα οποία πρέπει να είναι θετικά, αλλά να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε κυρίως για να βοηθήσουμε και τους νέους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζουμε πλήρως αυτό το ψήφισμα Όσο μεγάλες και αν είναι οι διαφορές μεταξύ ανθρώπων δεν επιτρέπεται να καταλήγουμε στην βία. Και δεν πρέπει να μειώνεται και το δικαίωμα βεβαίως να περιορίζουμε τον ελεύθερο λόγο. Αλλά βεβαίως υπάρχουν τα όρια του όταν καλούμε σε βία. Έτσι, όταν κάποιος με τα λόγια του καλεί σε άσκηση βίας είναι διαφορετική περίπτωση. Ε, ε, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν ε, Ολλανδοί δημαρχοί με συνοδεία αστυνομία στη δουλειά τους επειδή τους απειλούν. Είναι φρικτή κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ντονάτο Τόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ του ψηφίσματος αυτού και υπέβαλα μια τροπολογία για να ενισχύσουμε το σημείο 9. Το τμήμα αυτό αφορά εις το μίσος μέσω ανώνυμων μηνυμάτων στα, κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία μέσα πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνα από όσο τους επέτρεψαν να είναι τα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα, πρέπει να κάνουν περισσότερα τα κράτη-μέλη και ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι αυτό το ψήφισμα. Διότι μέσω ανώνυμων τέτοιων δημοσίευσεων εκφράζονται τα χαμηλότερα ανθρώπινα ένστικτα και όταν αυτό γίνεται ανωνύμως χρησιμοποιούν την πιο βίαιη ορολογία, την πιο ταπεινή ορολογία και ένας τέτοιος έλεγχος, ε, μάλλον μια τέτοια έκφραση μίσους ε, γίνεται με πολλούς τρόπους και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός που υπογράφει τα λεγόμενά του τουλάχιστον αναλαμβάνει την ευθύνη της άποψής του. νομίζω ότι πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα, Πρόεδρε, για το λόγο αυτό. Ο τελευταίος ομιλητής ε, είναι ο Γκαϊτάνο Αρμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για την απόσυρση της τροπολογίας ε, υπαριθμών 2 με το περιεχόμενο που καλούσαν όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους κομμάτων δηλαδή, αλλά και θεσμών, αποφεύγοντας ε, επιθετικούς όρους και όρους που εκφράζουν μίσους, παράλληλα υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα έκφρασης, ήταν η ίδια πρόταση που έκαναν και ο συνάδελφος Βόσνια και άλλοι Πολωνίοι συνάδελφοι όπως και ο κύριος Ανταμόβιτς που τον θυμόμαστε σήμερα αποσύρω λοιπόν τροπολογία και υποστηρίζω το ψήφισμα διότι η Ευρώπη θα πρέπει χάνουμε το μικρόφωνο του μιλητή την καταπολέμηση του, των μηνυμάτων μίσους. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος μετά την γενική αυτή συζήτηση. Α, όχι, ο κύριο ε, Σουνάιντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία να κάνω μια τροπολογία, μια πρόταση. Δεν έχουμε κάποιον εισηγητή, γι' αυτό είναι κάπω περίεργη η διαδικασία. Το θέμα μου είναι το σημείο 4. Στο σημείο 4 λέμε ξεκάθαρα πως με αφορμή την δολοφονία του κυρίου Άμπραμόβιτς λέμε ότι πολλοί δήμαρχοι που είναι εδώ πέρα σε αυτήν την αίθουσα είναι θύματα επιθέσεων λεκτικών αλλά και βίαιων πράξεων. Ε, πάρα πολύ βασικό αυτό. Υπάρχει μια τροπολογία τώρα της κυρίας Όνε να μιλήσει για μέλη της κοινωνίας των πολιτών είναι ε, σωστό αυτό, αλλά δεν ταιριάζει εδώ. Οπότε προτείνω το κείμενο της κυρίας Ωνέ να μπει ως χωριστή παράγραφος μετά το σημείο 6. Απλά το λέω για να το δούμε στην διάρκεια της ε, ψηφοφορίας. Ε, δεν ξέρω, η συντάκτης τι έχει να μας πει. Εγώ συμφωνώ ναι, και έτσι νομίζω θα ε, επιτευχθούν ε, και οι στόχοι μας. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν. Περνάμε. Περνούμε στις τροπολογίες και στην τροπολογία 4 μιλήσουμε για την τροπολογία του κυρίου Σνάιντερ. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αποσύρεται, όπως ακούσαμε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου Σνάιντερ για να έχουμε χωρισμό της ε, παραγράφου σε ένα σημείο το οποίο εκείνος υπέδειξε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4 έτσι όπως τροπολογήθηκε. Υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Όχι. Ο κύριος Τομά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ υπέβαλα την τροπολογία 6, αλλά έχω την πρόθεση να αποσύρω. Ίσως είναι καλύτερα να εστιαστούμε στην τροπολογία 5 και κατά την άποψή μου έχει το ίδιο περιεχόμενο. Αποσύρω λοιπόν την 6, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 6 αποσύρεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα με ομοφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνούμε τώρα στην ε, σύνηθε θέμα, θέματα που αφορούν τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία έστειλαν υποδείξει για διάφορα θέματα προ μελέτη. Δεν μπορέσαμε να τα επεξεργαστούμε όλα, είναι θέμα χρόνου. Η διάσκεψη των Προέδρων παίξε τρία θέματα που θα συζητήσουμε τώρα διαδοχικά. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα, ανάπτυξη σχέσεων με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Μολδαβίας. Χαιρετίζω το ότι το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνει στη μερίσια διάδειξη σήμερα, διότι είμαστε σε μόνιμη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Μολδαβίας διαμέσου της ε, δομής που έχουμε για την εταιρική σχέση με τις εταιρικές σχέσεις. Και όπως ξέρετε η Μολδαβία θα έχει την συμπροεδρία το 2022. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Μολδαβίας που είναι σήμερα μαζί μας και με την οποία μπόρεσα να συζητήσω την τρίτο απόγευμα να συζητήσω θέματα συνεργασίας με την Επιτροπή μας. Η συνεργασία αυτή γίνεται μέσω των εργασιών που έχουμε στην Επιτροπή ΣΥΒΕΞ ή με άλλα συγκεκριμένα γεγονότα όπως το Φόρμ για την Εφόρο Ανάπτυξη, την Γενική Συνέλευση για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες ή την Διάσκεψη Κορυφής στο Βουκουρέστι και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων και Περιφερειών. Θα ήθελα τώρα να δώσω στον συνάδελφο Αντριάν Τεμπάν το λόγο για να παρουσιάσει το σχετικό θέμα. Κύριε Τεμπάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως Αντιπρόεδρος θα ήθελα να σας πω με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Επιτροπή Περιφερειών να υποστηρίξει την ε, πορεία μας προς την Ευρώπη. Τα τελευταία 25 χρόνια η Μολδαβία έκανε σημαντικές προσπάθειες αποκέντρωσης και μπορούμε μετά από αυτές τις, με αυτές τις προσπάθειες να σας πούμε τι έχουμε κάνει, αλλαγές, τους ε, νομικής ε, τάξης για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη αυτονομία στις περιοχές. Επίσης, ε, βελτίωση των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών και φορολογική αποκέντρωση. Τα τελευταία χρόνια όταν μιλούμε για τοπική ανεξαρτησία έχουμε εγκρίνει διάφορες νομοθετικές πράξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την μεταρρύθμιση της δημόσιας δίκησης. Το 2016 έγιναν μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο πάρα πολύ σημαντικές και θεωρήθηκαν θετικές. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις μεταρρυθμίσεις για την τοπική δημοκρατία και για την ενίσχυση των δεσμεύσεων που προανέφερα. Όσον αφορά την πρόοδο σε επίπεδο τοπικού επίπεδου δημοκρατίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά είναι επιτυχής. Είμαστε μέλος της ε, εταιρικής σχέσης των ανατολικών χωρών. Πρέπει να πω ότι κάποιες φιλελεύθερες τάσεις παρουσιάστηκαν σε επίπεδο τοπικής ε, αυτοδιοίκησης και διακυβέρνησης. Στην Μολδαβία οι τοπικές αρχές όμως δεν έχουν αρκετή εξουσία ώστε να μπορέσουν να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να κάνουν σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορούν πάντα να το κατορθώσουν. Άρα θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία ώστε να μπορέσουν οι τοπικές αρχές να συμμετέχουν περισσότερο σε τοπικές δράσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποκέντρωσης σε μια χώρα στην οποία υπήρχε πλήρης ε, ε, κεντρικοποίηση και υπερσυγκεντρωτισμό στην κεντρική εξουσία την εποχή της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Άρα πρέπει να καταβληθούν για αυτό το θέμα ακόμη περισσότερες προσπάθειες. Η αποκέντρωση σε τοπικό επίπεδο κάποια στιγμή σταμάτησε και η το κυβερνών κόμμα είναι μάλλον κατά της αποκέντρωσης. Στα πλαίσια της Κορλεάπ, οι τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές είναι υπέρ του να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Στα πλαίσια αυτού του φόρουμ μπορούν να τονιστούν περισσότερο οι βέλτιστες πρακτικές και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερη δύναμη μετά από διαπραγματεύσεις στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα εξέφρασε την υποστήριξή του προς τις τοπικές αρχές στην Μολδαβία μέσω του ψηφίσματος του σχετικού και αυτό είναι κάτι το οποίο αναλάβαμε να μεταφέρουμε και στις αρχές μας. Ξέρουμε ότι θα πρέπει όλο και περισσότερο να ακολουθούμε τα αχνάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυρίως αυτό αφορά τα νέα παιδιά, τους νέους κάτω των 30, που πρέπει να συσφίξουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις δικές σας προσπάθειες μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα στην επόμενη θητεία να θεσπίσουμε μια ειδική ομάδα εργασίας για τις σχέσεις με τη Μολδαβία λαμβάνοντας υπόψη ποιες βήματα έχουν γίνει στην δική μας χώρα και στις υπόλοιπε χώρες της ε, Ανατολικής εταιρική Σχέσης και σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε άλλες παρατηρήσεις, άλλες παρεμβάσεις επί του σημείου αυτού της διατάξεως. Δεν έχει εγγραφεί κάποιος ομιλητής εδώ. Δεν βλέπω κάποιος να ζητάει το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Λέγοντας ότι θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση για την 25η επέτειο των τοπικών αρχών και του Συμβουλίου της Ευρώπης 26 και 27 Ιουνίου. Στο συνέδριο αυτό θα εξεταστεί το καθεστώς της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στην Ευρώπη ως πρόσθετος ε, μάλλον θα υπάρξει και ένας πρόσθετος διάλογος ακριβώς για την ε, πρόοδο των, ε, την κατάσταση και τις προοπτικές των τοπικών και περιφερειακών χώρων στην Μολδαβία. Περνώ στο δεύτερο θέμα σε αυτή την ενότητα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, που υποστηρίζουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη δημοσίευση από την Κομισιόν του εγγράφου για την βιώσιμη Ευρώπη από εδώ στο 2030. Η Επιτροπή μας συνεισέφερε με τρία μέλη, Αμπραμαβίτσιους, Μπίβερ και Μπόσμαν, μέσω της ε, πλατφόρμας υπό τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς, έγγραφο που τρία χρόνια μετά την υπογραφή του θεματολογίου για το 2030 έδωσε συστάσεις ε, για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να αντιμετωπίσουμε μάλλον τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ακόμα η Ευρώπη και για την επόμενη δεκαετία στα πλαίσια της βιωσίμου ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν ένα έγγραφο, μια πρώτη ανάλυση, πρώτη μελέτη της πρόοδου της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε συγκεκριμένες τάσεις ε, σχετικά με τον αντίκτυπο της ε, κλιματικής αλλαγής που θα πρέπει να, να, προσανατολιστούν προτού τα πράγματα ε, να μην είναι πλέον αναστρέψιμα. Θα δώσω τώρα στον κύριο Ρώσα Μπαλας Τόρρες, ο οποίος επρότεινε το θέμα. Την κυρία Τόρρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητούμε σήμερα μέσω της ηγεσία που παρήχε και η Επιτροπή των Περιφερειών για την βιώσιμη ανάπτυξη αυτή την εβδομάδα Δευτέρα και Τρίτη. Οι τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές που είναι πολύ κοντά στον πολίτη θα πρέπει να προσπαθήσουν ε, για την ανάπτυξη και την ατομική και των κοινωνιών και οικονομιών μας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια από τις πιο σημαντικές μας ευθύνες ως τοπική διοίκηση και αυτό θα πρέπει να γίνει με συνέπεια το θεματολόγιο 2030 του στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όλα αυτά θα πρέπει να συγκλίνουν σε μέσα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε τις δημόσιες πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να είναι συνεπείς και να αναπτυχθούν στο έδαφος ε, υπό την αρμοδιότητά μας ε, ως Παροχή υπηρεσιών, υπολίτιμων ε, υπηρεσιών προ του πολίτε. Αυτό θα, γίνει, θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τι ενεργειακέ πολιτικές και τις πολιτικές αναβιομηχάνησης. Όπως προσπαθούμε να κάνουμε και στη δική μου περιφέρεια στην Εξτρεμαδούρα και σε πλαίσια ε, διεθνού ε, συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να ευθεγραμμιστούμε λοιπόν ε, στις συστάσεις ε, των στόχων βιωσίμου ανάπτυξη ε, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας προκειμένου να επανέλθουμε σε μια πιο άμεση σχέση με σημαντικά τμήματα της κοινωνίας. Αυτό περνάει από μια τάση, μια κατεύθυνση όπου όλοι θα μπορούν να αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά το οποίο θα μας επιτρέψει και να κερδίσουμε νέα γνώση, να σωρεύσουμε νέα γνώση και να ανταλλάξουμε ε, γνώση με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε συνεργασία με τους πανεπιστημιακούς φορείς και τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα, το ίδιο ιδίωμα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ένα βιώσιμο μέσο ώστε να έχουμε μια νέα ε, ε, σύμβαση κοινωνική στις 26 Μαΐου οι πολίτες ε, θα κληθούν να ψηφίσουν και μεταξύ αυτών και νεαρότατοι πολίτες οι οποίες δεν έχουν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν. Νέοι δηλαδή που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ε, και στην ε, οικονομία και στην ε, τεχνολογία και με συγκεκριμένες κρίσεις τοπικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζουμε και στη δική μας περιφέρεια. Νέοι που θέλουν πάνω απ' όλα να συμμετάσχουν και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένας τρόπος για αυτούς να αισθάνονται πιο κοντά στα κέντρα λήψεως απόφασης και γι' αυτό συνάδελφοι και από τις δικές μας τοπικές διοικήσεις θα πρέπει να αναπτύξουμε διαδικασίες που θα επιτρέπουν να ακούμε τους πολίτες και να υλοποιούμε τις ιδέες τους σε πραγματικότητα. Γιατί οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι ίδιοι οι πολίτες, η ίδια η κοινωνία. Ολοκληρώνω. Το θεματολόγιο 2030 θα πρέπει να είναι εκείνο το μέσο που θα μας επιτρέψει να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, να μην ξεχάσουμε κανέναν, και το θεματολόγιο αυτό θα πρέπει να το υλοποιήσουμε επί τη βάση του νέου αυτού ε, συμφώνου ώστε οι πολίτες να μην αισθάνονται πλέον απομακρυσμένοι από το ευρωπαϊκό όραμα και έργο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι σαφές και στα βασικά ψηφίσματα και στους στόχους ε, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών νομοθετών. Αλλά βεβαίως Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και στο τοπικό επίπεδο. Και έχουμε τους στόχους ε, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχει αναλλακτική σε αυτά τα πράγματα. Όταν μιλάμε τώρα για το τοπικό επίπεδο θα πρέπει οι πόλεις μας ε, να γίνουν πιο ε, περιληπτικές ε, μέσω έργων που θα θέσουν ακριβώς τις βάσεις για τέτοια βιώσιμη ανάπτυξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βεβαίω ένα σημείο που εστιάζουν αυτές οι δραστηριότητες και πρέπει να υπάρξει και ένα επιχειρηματικό πνεύμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή οι τοπικές αρχές να τα καθορίζουν αυτά ε, παράλληλα με τις εθνικές ε, αρχές και τις ευρωπαϊκές αρχές. τη ε, φάση της εφαρμογής επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, φορολογικές και από πλευράς προσωπικού. Ως εκπρόσωπος λοιπόν ε, κροατικών ΟΤΑ θα ήθελα να είμαι τέρος. Σας ευχαριστώ Λουρή και Χιλόχ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Κοιτάξτε και μας μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτοί οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2030 έχουμε την ευκαιρία ε, να δούμε αυτούς 17 στόχους για έναν καλύτερο κόσμο από κοινού, να τους εφαρμόσουμε και όπως ήδη αναφέρθηκε το θέμα είναι η καταπολέμηση της στόχιας, οι ανισότητες, προστασία του περιβάλλοντος, δικαιώματα των γυναικών, εκπαίδευση. Εμείς ε, στην Βρέμη απευθυνόμαστε με απλή γλώσσα στους πολίτες ε, και τους δίνουμε τη δυνατότητα να λάβουν μέρος ε, και τον Μάρτιο είχαμε αυτήν την δεύτερη διάσκεψη συνεργασίας των πόλεων είναι σημαντικό λοιπόν να ανταλλάσσουμε απόψεις ε, τα καλά παραδείγματα που έχουμε για τους διάφορους στόχους. Η Βρέμη βεβαίως ε, εμπλέκεται στον τομέα του δικαίου εμπορίου των κοινωνικών στόχων και βεβαίως ε, χαιρόμουν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να σκεφτούμε από κοινού πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ράνιτς έχει τώρα τον λόγο. Σας ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τρει σημαντικού στόχου που πρέπει να θέσουμε για την ενέργεια. Την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας, ε, παγκόσμια ηγεσία στις ανανεώσιμες και η χρήση καθαρής ενέργειας για όλους τους πολίτες μας. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Το σύμφωνο των δημάρχων με εκατοντάδες ε, ε, ε τέτοιες ε, τοπικές αρχές που έχουν δεσμευτεί και υπάρχει ο ρόλος ε, των δημάρχων που τονίζουν την χρήση των ανανεώσιμων πηγών. Η ΟΤΑ λοιπόν σε πολλά κράτη-μέλη είναι ένα βήμα α, μπροστά από τα κράτη-μέλη Έχουμε λοιπόν κάποια τοπικά βήματα που έχουν γίνει και έχει αναπτυχθεί μια τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να τονίσω την σημασία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και επίσης την ανάγκη του να αυξηθεί η ορατότητα των δράσεων αυτών ως προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω ότι οι χώρες οι οποίες λειτουργεί καλύτερα το σύστημα αυτό είναι πολύ καλά παραδείγματα γιατί έτσι επηρεάζονται όλες οι πτυχές της ζωής σε τοπικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Μακάρθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μας ακριβώς το ότι συνεργάζεται η Επιτροπή των Περιφερειών για τους στόχους αυτούς. Βεβαίως έχουμε τρία-τέσσερα χρόνια να δούμε ε, εδώ πέρα εκπροσώπους του ΟΗΕ. Είναι, είναι ένα βάρος λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει εμείς ε, να σηκώσουμε, να ανταποκριθούμε στην ε, νέα αστική ατζέντα του ΟΗΕ. Πρέπει να ανταποκριθούμε στους στόχους της αστικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συνδέσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, στον ΟΗΕ και στο Φόρουμ Υψηλού Πολιτικού Επιπέδου με το πι δέλτα πι. Συνολικά λοιπόν κύριε Πρόεδρε πρέπει να κινητοποιηθούμε περισσότερο όσον αφορά την ανάπτυξη, να είμαστε περισσότερο εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ανάπτυξη των στόχων της χιλιετίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε <clears throat> και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να τονίσω τους στόχους 14-15 δηλαδή <clears throat> για, τον, για το χερσαίο και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Σε αυτό τον πράσινο και γαλάζιο δηλαδή κόσμο που αποκαλούμε τον πλανήτη μας. Πρέπει να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα που έχει άμεση σχέση με το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και τους στόχους του 2030. <clears throat> Μόνο σεβόμενοι αυτό το οικοσύστημα θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία και μια ανταγωνιστική οικονομία που να βασίζεται στη γνώση. Είχα την τιμή να εκπροσωπώ την Επιτροπή των Περιφερειών στην COP14 των Ηνωμένων Εθνών <clears throat> για την βιοπικιλότητα τον περασμένο Νοέμβριο και με μεγάλη χαρά μπορώ να σας ανακοινώσω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών αναγνωρίζεται ως διεθνής φορέας στα θέματα της βιοπικιλότητας και στην προστασία της. Νομίζω ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, εντός του πλαισίου των πολιτικών των σημερινών και των μελλοντικών για την προστασία της βιοποικιλότητας. Έχοντας δουλέψει για ένα χρόνο στην πλατφόρμα των ενδιαφερομένων ε, μερών για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για τους στόχους πάνω από όλα όπως έλεγα 14 και 15 σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για να ολοκληρώσω αγαπητοί φίλοι, Πραγματικά ενθαρρύνω όλους και όλες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να αναλάβουμε τις ε, ε, ευθύνες μας για την βιώσιμη ανάπτυξη και την βιοποικιλότητα. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε τώρα την συζήτηση με, τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Μάρκουλα. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ε, τοποθετήσεις τους ε, και τη συνεισφορά τους. Έχουμε ακούσει σημαντικά μηνύματα για τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών που είναι σημαντικός αλλά μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικός και σε αυτό πρέπει να εστιαστούμε ε, για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Και η σημασία μας είναι παράλληλη με το πόσο Ενεργεί είναι οι πόλεις και οι περιφέρειες εστιαζόμενοι στις, στη ζωή των επιχειρήσεων, των πανεπιστημιακών φορέων, της έρευνας εκτός των διοικητικών υποθέσεων. Είχα την ε, τιμή να συμμετάσχω μαζί με, τον, ε, με την ε, κυρία Χέρτελη όπου εστιαστήκαμε στις, ε, στους στόχους βιωσίμου ανάπτυξης μαζί με εκατοντάδες ε, εκπροσώπους επιχειρήσεων και δήμων για να δημιουργήσουμε κοινέ δράσεις, να σχεδιάσουμε κοινέ δράσεις ώστε η ε, Δήμη να είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την προσπάθεια αυτή. Και αυτό κάνουμε και στην Επιτροπή των Περιφερειών, τονίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ξεκινήσει πλέον ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την ηγεσία των Δήμων και των Πόλεων ή στην προσπάθεια ε, ε, για τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης, δεσμεύοντας και σημαντικούς πόρους σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτή τη δουλειά και σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να χρειαστούμε την ενεργό συμμετοχή όλων και θα πρέπει να είμαστε πρέσβεις ε, παγκοσμίω ε, τη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο κύριος Αμπραμοβίτης και η κυρία Χέρτελη προετοιμάζουν το πλαίσιο αυτό της προσπάθειας ε, μέσω της οποίας θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Επιτροπή των Περιφερειών και το σημερινό και τον μελλοντικό. Σας ευχαριστώ. Όπως το είπε και ο κύριος Μάρκουλα θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό κατά την Ολομέλεια του Ιουνίου με τις ε, δύο γνωμοδοτήσεις που ε, θα υποβληθούν για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Φτάνουμε τώρα στην τρίτη θεματική της ενότητος, τον εδαφικό δηλαδή αντίκτυπο του Brexit. που σήμερα είναι και της απολύτου επικαιρότητος ε, δεδομένης της ε, επίσκεψης της ε, Πρωθυπουργού ή στις Βρυξέλλες. Η απειλή λοιπόν της άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου γίνεται όλο και πιο έντονη πλησιάζοντας στην καταληκτική ημερομηνία «The clock is ticking» που λέμε και στα ελληνικά. Επομένως εντείνουμε και τις προσπάθειες προετοιμασίας μας. Ε, η Κομισιόν έχει οθετήσει ένα έκτακτο σχέδιο ανάγκης ε, με διάφορες πρωτοβουλίες για να αποφευχθούν προβλήματα στις ε, αέριες μεταφορές, τελωνιακές δυσκολίες, στην εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων, πρόβλημα αντιμετώπισης στα σύνορα της Βορείου Ιρλανδίας, και να αντισταθμίσουμε τον αντέκτημο που θα είχε ε, μια τέτοια αποχώρηση και στην Αλία όπως και στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Βέβαια ε, ένα Brexit άτακτο θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και όπως έχει δείξει συγκεκριμένες μελέτες θα είναι ασύμετρος αυτός ο αντίκτυπος σε κάποιες περιφέρειες πολύ πιο έντονα από τις άλλες. Αυτό φάνηκε και στο ψήφισμα του Μαρτίου του 17 και του Μαΐου 18 με σειρά ανησυχιών που συνελέχθησαν από τον επικεφαλής διαπραγματευτή για τις Ευρωπαϊκής Ένωση τον κύριο Μπαχνιέ και που είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στην περασμένη Ολομέλεια. Θα δώσω το, το λόγο στον κύριο Ντεκόστερ, ο οποίος εισήγαγε το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι από μια περιοχή, τα Old House, που πάντα κυνηγούσε ένα όνειρο. Το όνειρο να μπορέσει να περάσει την μάχη όχι πλέον ως εμπόδιο, αλλά ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας. 40 χιλιόμετρα μόνο. Πρόκειται λοιπόν τώρα για μία ε, μέτρηση αντίστροφα της απόστασης που μας χωρίζει. Θέλουμε όλο και πιο, όσο και πιο γρήγορα να φτάσουμε εκεί. Αλλά την ε, απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας τη σεβόμαστε. Απόφαση ενός λαού ολόκληρου, αλλά παράδοξη αν βρούμε ποιοι είναι οι δεσμοί που μας συνδέουν εμάς στην περιοχή Όντεφχός και τους φίλους μας της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης πρέπει να πω ότι είμαστε μπροστά μια παράδοξη κατάσταση με τον ε, κύριο αντικειμενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα πρώτα απ' όλα. Τα σύνορα που όπως υπενθύμησα στην ιστορία που σας είπα πρέπει να είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ των λαών μας. Το Brexit είναι ουσιαδού σημασία γεγονό στην ιστορία μας και θα είμαστε όλοι χαμένοι από αυτήν την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλη της η επικράτεια και το ίδιο το ε, η Μεγάλη Βρετανία. Πραγματικά πρέπει να πω με άλλους 21 συναδέλφους μου ε, από τον Ιανουάριο πέρσι και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αντιπροέδρους αυτής της ε, ε διαπεριφερειακής ομάδας σε κάθε ολομέλεια μελετούμε τις πιθανές συνέπειες του Brexit για θέματα ενέργειας κυκλοφορίας, ε, ε, παράκτηων μεταφορών, ε, αλλίες κτλ. Και σήμερα το πρωί και έναν από τους συνεργάτες του κυρίου Μπαρνιέ. Ξέρουμε ότι με την ενίσχυση όλων των ελέγχων φυτοϊγειονομικών, τελωνιακών διότι ξέρουμε ότι δεν έχουν ληφθεί τα ανάλογα μέτρα, θα υπάρχουν ε, άγνωστοι πάρα πολλοί χ για όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και τις μιμίες που οι οποίε δούλεψαν με αγαστή συνεργασία στα πλαίσια του γίου συντονισμού τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι η Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να συνοδεύσει περιφέρειες της Ευρώπης οι οποίες θα υποστούν τις περισσότερες συνέπειες. Πρώτα απ' όλα, όντας ακόμη πιο παρούσα η Επιτροπή μας στις μελλοντικέ συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να αντιγράψουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έστειλε έναν συνάδελφο να παρακολουθήσει τις ε, συζητήσεις και να συνοδεύει όλες τις συζητήσεις που γίνονται. Και επίσης να ζητήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν στις περιφέρειες που προανέφερα και στις περιοχές να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτή την κατάσταση. Όπως είχε γίνει παλιά με τις ε, ε παραμεθόριες περιοχές, αν μπορώ να τις πω έτσι, προς την Ανατολική Ευρώπη, όταν ε, πριν να γίνει η τελευταία ε, διεύρυνση. Ο κύριος Ζουλιό και ο κύριος ε, Μάνια έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα μία τέτοιου είδους πρόταση και πιστεύω ότι στην σχετική τροπολογία 45 λέγεται ότι θα πρέπει να ευρεθούν πάρα πολλές ε, λύσεις για να βοηθηθούν οι όμερες περιοχές προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση και να υποστηρίξουμε μέσω των Ευρωβουλευτών μας την τροπολογία αυτή να περάσει την επόμενη εβδομάδα στη Στρασβούργο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Έχουμε την ε, τρέλα του Brexit και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ξεκινήσω με το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης μετά από 15 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων που σωστά περιγράφτηκαν από τον Γενικό Γραμματέα της Κομισιόν ως δημοκρατικό αριστούργημα. Ένα συμβασμός και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως ένα σχέδιο συμφωνίας, το οποίο συμφώνησαν και οι δύο πλευρές τον Νοέμβριο πέρσι. Η Επιτροπή των ε, Περιφερειών ε, είναι πολύ δραστήρια στην συζήτηση του Brexit και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία δεδομένου του ότι οι συνέπειε του Brexit θα γίνουν αισθητέ σε τοπικό επίπεδο. Μία συζήτηση την οποία ξεκινήσατε εσεί, ε, κύριε Πρόεδρε. Οι πολιτικές ομάδες, ε, η ομάδα υπό την ηγεσία του κύριου Φρανσουά Ντεκόστερ. Επίσης ε, θα θέλαμε να αναφέρουμε ιδιαίτερα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ που έκανε επίσης αυτόν τον την μελέτη περιφερειακών αντικτύπων ε, και βεβαίως οι αντίκτυποι διαφέρουν, όλες οι περιφέρειες ε, θα επηρεαστούν, όλες οι περιφέρειες που εκπροσωπούνται σε αυτήν την αίθουσα. Βεβαίως πιο κοντινές, ε, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία και βεβαίως και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά Αυτό το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο είναι η ειρήνη στην νήσο της Ιρλανδίας που είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια η οποία βεβαίω δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν είχαμε 30 χρόνια φρικτής βίας. Ε, μια ειρήνη λοιπόν εύθραυστη. Υπάρχουν ακόμα εντάσεις, διχασμένες ε, κοινότητες, παραστρατιωτικοί που είναι ενεργοί. Εξού και το περίφημο αυτό το backstop το οποίο εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει ε, σκληρό σύνορο στην Ιρλανδία αλλά θα προστατεύει και την ε, ενιαία κοινή αγορά. Την τρίτη που μας πέρασε είδαμε την Βρετανίδα Πρωθυπουργό να υπαναχωρεί από αυτήν την συμφωνημένη θέση και ε, ε η μεταβολή αυτή της Βρετανίδας Πρωθυπουργού ενισχύει ακριβώς την ανάγκη του να υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για να αποφευχθούν τα σκληρά λεγόμενα σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν, εάν υπάρξουν τεχνικές λύσεις στο μέλλον, να ξαναδούμε το θέμα τότε. Για όλους λοιπόν εντός της ε, αιθούσης, το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε μια έφτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου ή να υπογράψουμε το σχέδιο συμφωνίας που είναι προς το συμφέρον κάθε περιφέρειας εντός αυτής της αιθούσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται το κατάλογο των ομιλητών διότι θα πρέπει λίγο να σεβαστούμε το χρόνο που έχουμε στην ε, διαθέσή μας. Ο κύριος Όχτα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάλυση που έγινε για την διαδικασία αποχώρησης που χαρακτηρίστηκε ως παράδοξη για τον Brexit και θα πρέπει να επισημάνουμε κάποιους ε, κινδύνους που έχει για τη δημοκρατία το θέμα αυτό, αντίθετα με την θέληση των λαών. Η άτακτη αποχώρηση τη μεγάλη Βρετανία, τη στιγμή στην οποία βλέπουμε να μαζεύονται σύννεφα πάνω από την παγκόσμια οικονομία είναι ένα μεγάλο κίνδυνο για όλου. Εκτό από τα πολιτικά προβλήματα για την ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κοινωνικέ και οικονομικέ συνέπειε μεγάλη σοβαρότητα. Γι' αυτό καταλόγουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμφωνία που θα γίνει μεταξύ μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό. Αν ξαναρχίσουν διαπραγματεύσει αν υπάρχουν αμφιβολίες για την βούληση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μεγάλη Βρετανίας να προχωρήσουμε θα είναι κάτι επικίνδυνο και για μας και για την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να σα πω επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της μεγάλη Βρετανίας ο γεωστρατηγικό για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Υπογραμμίζω είναι πολύ σημαντική η θέση της Μεγάλης Βρετανίας και κατά τη διάρκεια της επίτευξης του Brexit και μετά. Γι' αυτό εκφράζουμε την ευχή η επίσκεψη της κυρίας ε, ε, Μέη στις Βρυξέλλες να είναι καρποφόρος και θετική. Ευχαριστώ. ο ομιλητή, ο συνάδελφος Ρουμπά. Ε, I would just like to mention that Ήθελα απλά να πω πως ε, έχει μεγάλη σημασία η περιφέρεια Μπράτισλάβας για την αυτοκίνητο βιομηχανία. Η Σλοβακία μετά τη μεταρρύθμιση της βαριάς στρατιωτικής βιομηχανίας έγινε η χώρα με την υψηλότερη παραγωγή αυτοκινήτων ε, αναλογικά με τον πληθυσμό. Ε, καθώς μετακινήθηκαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε χώρες με φτηνότερη εργασία μετά τη διεύρυνση του 2004 και πρόκειται για ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της ε, Σλοβακίας και βεβαίω ε, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων. Η Σλοβακία δεν έχει βεβαίως εγχώριους κατασκευαστές, έχουμε τέσσερις μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες εξαρτώμεθα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα κεντρικά οι περιφέρειές της λοιπόν αντιμετωπίζουν τους κινδύνους από αυτές τις αποφάσεις. Στην Σλοβακία έχουμε τη Volkswagen, ε, ναι, την Peugeot, την Kia και την Jaguar Land Rover, την αγγλοϊνδική εταιρεία που ξεκίνησε και αυτή πρόσφατα την παραγωγή. Ανησυχούμε πάρα πολύ για το πώς θα μας επηρεάσει το Brexit, τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 53 μέρε πριν το Brexit έχουμε ακόμα μεγάλες αβεβαιότητες. Ελπίζουμε να υπάρξει μια ικανοποιητική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και ε, να βρεθεί σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στένσον. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι από μια μεθοριακή περιοχή της Ιρλανδίας ε, και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον Brexit. Δεν εμπιστευόμαστε πλέον τους Βρετανούς ότι θα φύγουν ε, έφτακτα από την Ένωση. Και να ρωτήσω εδώ πέρα τους Μπρεξιτικούς, ε, ξέρετε τι θέλετε τελικά, πρέπει να πείτε τι θέλετε να γίνει. Και πρέπει να σταματήσετε να α, λέτε ψέματα για την δικλίδα ασφαλής. Απλά θέλουμε να μην υπάρχουν σκληρά σύνορα στην Ιρλανδία. Για το Brexit μας είπαν ότι θα είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Μα ήταν τόσο εύκολη δεν θα χρειαζόμασταν αυτήν την εγγύηση στην Ιρλανδία. Το θέμα δεν θα πρέπει να είναι οι προνομιούχοι στην ε, Βρετανική Βουλή αλλά το τι γίνεται στην περιοχή μας, ειδικά τη δικιά μας, την μεθοριακή. Ε, μαθητές που ίσως χρειαστεί να αλλάξουν σχολείο, άνθρωποι που δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Και πολλοί άνθρωποι που θα χάσουν τις δουλειές τους, άρρωστοι, που δεν θα έχουν πρόσβαση στο κοντινότερο νοσοκομείο. Και βεβαίως ε, οι κοινότητες ε, που ίσως χωριστούν πάλι από τα σύνορα. Γνωρίζουμε λοιπόν τις συνέπειες που θα έχει ένα σκληρό σύνορο στην Ιρλανδία και κανεί δεν θέλει να επιστρέψει στη βία του παρελθόντο. Γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε την δικλίδα ασφαλεία. Ω αγρότη δε, εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι αυτό θα βλάψει την γεωργία μας καθώς έχουμε οικοδομήσει και ένα εμπορικό σήμα ε, Ιρλανδικό και ως πατέρας ε, δεν θέλω να δώσω στα παιδιά μου λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι είχα εγώ και ως ερετός Πραγματικά δεν θέλω να σκέφτομαι το τι σημαίνει αυτό για τις μεθοριακές κοινότητες. Πρέπει επιτέλους οι Βρεξιτικοί να σταματήσουν να κατηγορούν τους Ιρλανδούς και τις Βρυξέλλες. Να κοιτάξετε στον καθρέφτη και να κατηγορήσετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Καλαμπουίκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι λογικά όλοι σεβόμαστε την απόφαση του λαού της Μεγάλης Βρετανίας. Εκ των υστέρων όμως μας φαίνεται ότι είναι λανθασμένη απόφαση που θα δημιουργήσει σοβαρότητα προβλήματα στην Ευρώπη, αλλά κατά κύριο λόγο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ είμαι από μία περιοχή, από τη Βαλένθια, που για μας είναι αυτό πρωταρχική σημασία, Αλλά όπως είπε και ο κύριος Μπαρνιέ, τον οποίο είδαμε πολλές φορές, θέλουμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό που θέλουμε είναι κυρίω να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των πολιτών. Έχουμε περίπου 100 χιλιάδες ε, Βρετανούς που ζουν στην Ισπανία και 30.000 Ισπανοί ζουν στην Μεγάλη Βρετανία. Θέλουμε λοιπόν να, να μην σταματήσουν να έχουν τα δικαιώματα που έχει κάθε πολίτης στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και είμαστε αλληλέγγυοι επίσης ε, προς όλα τα στοιχεία που αφορούν την ερευτική διαδικασία και την Ιρλανδία, διότι αφορούν όλους τους πολίτες. Αλλά προφανώς θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη τους πολίτες, τα δικαιώματά τους, αλλά και τους διάφορους ε, τομείς, τον ε, αγροτικό, τον ε, διατροφικό, τις βιομηχανίες και πρέπει να πούμε ότι για μας κυρίως τα τρία εκατομμύρια Βρετανοί που έρχονται στην περιοχή μου κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, τα θέματα Συνδεσιμότητα διασύνδεση για τι εναέριε ε, μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντικά. Α σταματήσει αυτή η τρέλα, α καταλήξουν όλοι οι ενεχόμενοι σε μία λογική συμφωνία διότι αυτό το αποφάσισαν οι Βρετανοί. Λυπούμαστε που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αλλά θα πρέπει να βρεθεί η τελική λύση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κούπερ. Hello. Uh, Φίλοι Ευρωπαίοι, είναι η τελευταία ολομέλεια για τη Μεγάλη Βρετανία, ίσως, ίσως. Και αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Το Brexit ή το no Brexit, ό,τι και να συμβεί, ακόμη είμαστε ενωμένοι με πολλαπλούς τρόπους προς το ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ που ασχολούμαι με την ε, κλιματική αλλαγή στα πλαίσια της Επιτροπής Περιφερειών, ξέρω ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Παρακολουθούμε στα πλαίσια της ΚΑΠ21 ε, με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και ξέρουμε ότι έχουμε τέτοια πολλά, πολλά παραδείγματα. Λένε εδώ οι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση. Εγώ δεν σέβομαι την απόφαση του δημοψηφίσματος που βάθηκε σε ε, αυτά τα οποία προέβαλαν ως ιδέες ο Φάρατζ, ο, ο Μπόρις Τζόνσον και άλλοι. Βασιζόμενοι σε ψέματα, σε αυταπάτες, σε οτιδήποτε μπορούσαν να κάνουν για να εξαπατήσουν το λαό μας και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, σε αυτό το μπέρδεμα. Δεν τη σέβομαι την απόφασή τους. Και τώρα ξέρουμε ότι 56% των πολιτών μας θα ήθελα να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματική, πραγματικά πάρα πολλοί αισθάνονται ότι τους έχουν εγκαταλείψει. Ξέρουμε ποια είναι τα πολλαπλά ωφέλη που έχουμε. Η εκστρατεία αυτή, η οποία ίσως χρηματοδοτήθηκε από κάποιες σκοτεινές δυνάμεις, για να το πω απλά, So if we do leave the EU, there is a responsibility on us who go back. Από δυνάμεις μεταξύ άλλων για να εξασφαλιστεί το ότι ε, ό,τι έγινε δεν έγινε μόνο από αυτούς αλλά με κοινικό τρόπο από άλλους είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Θα πρέπει να προσφέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο την πολιτική της ελπίδας, του να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ολοκάνουμε θετικά για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε κατά αυτών που είναι υπέρ του Brexit. President, and uh, I'm sure that the majority, if not everybody. Είμαι σίγουρος πως η πλειοψηφία θα συμφωνούσε με την αρχική σας δήλωση πως το Brexit και ένα σκληρό Brexit όπως λέγεται χωρίς συμφωνία θα στείλει πραγματικά τεράστιους κραδασμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό όμως. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δήμοι, κάποιες περιοχές, κάποιες περιφέρειες η οικονομία των οποίων θα υποφέρει πολύ. Και η συνέπεια αυτού βεβαίως ε, είναι κάτι το οποίο θα νιώσουν οι πολίτες της Ευρώπης. Οι πολίτες οι οποίοι ε, είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Το Brexit θα επηρεάσει το πώς ταξιδεύουμε. Θα επηρεάσει τα πολιτιστικά μας ενδιαφέροντα. Το πώς γίνεται η έρευνα. Όλα αυτά κινδυνεύουν. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ πέρα και σκέφτομαι ένα τμήμα της κοινότητας Ευρώπης. Οι ναι. νέοι. Είμαι σίγουρος ότι αν γινόταν ένα ψήφισμα αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 70-80%, 90% των νέων θα ψήφιζαν να, για να μείνουν στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη που έχουμε σήμερα. Αλλά βεβαίως το μέλλον τους δεν είναι ένα μέλλον εθνών κρατών, αλλά μια ενωμένη Ευρώπης. Και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Φρανσουά Ντεκόστερ. Για ένα αστιάκι, αν θέλετε. Ένα αεροπλάνο που πετάει α, στους ουρανούς με μια ευρωπαϊκή σημαία στην ουρά και δύο άνθρωποι στέκονται στην ανοιχτή πόρτα. Συγγνώμη, λέει ο ένας. Ε, μήπως να παίρνατε και ένα λεξίτο το βγαίνοντας και ο άλλο απαντάει ε, όχι σας ευχαριστώ, η σημαία φτάνει και η σημαία είναι η Βρετανική βεβαίως. Συνάδελφοι, δεν μπορεί αυτό να είναι το μέλλον τη Ευρώπης. Δεν μπορούμε να τυλιγόμαστε στις σημαίες. Έτσι θα καταστρέψουμε τα όσα έχουμε οικοδομήσει τόσα χρόνια. Υπάρχουν α, πολύ περισσότερα πράγματα που κινδυνεύουν από το εμπόριο που αναφέρουμε. Η διάλυση της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά γιατί ο εθνικισμός αυξάνεται και το Brexit είναι μια μορφή αυτού του εθνικισμού. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue Sayed ο κύριος Σαγιέτ Μπίταν Νεύ. Η κυρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος επί των 27 όπως και επί της Ιρλανδίας. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον Μπελφάστ, γνωρίζω πόσο έχει επηρεάσει όλη η προηγούμενη ε, εμπόλεμη κατάσταση, οι συγκρούσεις ε, των προηγούμενων δεκαετιών. Δεν θα ήθελα καθόλου να επιστρέψουμε σε αυτές και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό τόπος στον παράδεισο και όχι στην κόλαση για αυτός που θα συνεισφέρουν σε μία λύση. Αφήνω την, τα, τις θέσεις στην κόλαση για τα διάφορα ρωσικά bots και άλλα, λέει ο Μιλήτρια. Εγώ πάντως ήθελα σήμερα να ζητήσω από όλους ως ο Αλίδα να κρατήσετε την πόρτα ανοιχτή, να διατηρήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Εμείς γνωρίζουμε ότι ήδη οι Ηνωμένε Πολιτείες και ο Καναδάς έχει ε, έχουν τοποθετήσει δασμού ε, στη χαλιβουργία μα και το ίδιο θα μα συμβεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον αποχωρήσουμε και το απέφχομαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο και, για, και το ίδιο είπε και ο δικός μας ε, πολιτικό ηγέτη ότι δεν πρέπει να κλείσουμε κάποια δυνατότητα, θέλουμε να διατηρήσουμε ό,τι και να γίνει μια θετική σχέση με όλου. Μιλήσαμε για τους νέους, μιλήσαμε για το πώς αυτό θα επηρεάσει το δικό τους μέλλον, θα επηρεάσει το μέλλον όλων μας με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, θα ήθελα πραγματικά να πω σε όλους και να βεβαιώσω άπαντες ότι είμαστε εδώ και θα είμαστε με θετικό πνεύμα πάντοτε για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Bentley, παρακαλώ τώρα. Bentley. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι νέο μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και είναι ίσως η πρώτη φορά που μιλώ στην Ολομέλεια και μπορεί και να είναι και η τελευταία. Ήθελα πάντως ε, να πω δύο λόγια για τα περιφερειακά και τοπικά συμβούλια, τοπικές αρχές δηλαδή, στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ως τοπική φορείς ένα διάλογο με την Βρετανική κυβέρνηση και μάλιστα εγώ ηγήθηκα μιας ε, ε, task force για την συζήτηση αυτή, τη διεξαγωγή της συζήτησης. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νομικών διατάξεων της νομοθεσίας ε, περνάει από τις τοπικές και περιβαλλικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν πρακτικός αντίκτυπος για τη δημόσια υγεία, για την ασφάλεια των τροφίμων για το περιβάλλον, όλα αυτά που δεν αναφέρονται μέσα σε όλο αυτό το πάθος της συζήτησης που είναι αντιληπτό, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε για να διασαβαλίσουμε τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν με γαλήνιο τρόπο, με ψύχρεμο τρόπο. Εμείς προσπαθούμε να συζητήσουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος επί των πολιτών και της οικονομίας. Γιατί το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, οι πολίτε, η δική του καθημερινή ζωή, η ευζοία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε στην όλη αυτή διαδικασία να μην υπάρξει αρνητικό αντίκτυπος. Όπως είπατε και εσείς ε, Πρόεδρε, θα πρέπει να αφού αποχωρήσουμε στις 29 Μαρτίου ή όποτε να διατηρήσουμε ένα διάλογο με την ε, Επιτροπή των Περιφερειών εγώ γνωρίζω ότι είμαστε πιο κοντά στον πολίτη από οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό κρατικό φορέα. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσουμε επιτυχώς και ομαλά τη διαδικασία αυτή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας ευχαριστώ. Χριστόφ Γουιόν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι το Brexit έχει αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταστροφικές για τη Μεγάλη Βρετανία. Ο καλύτερος τρόπος να απαφευθούν οι αρνητικές επιπτώσεις είναι να μην έχουμε Brexit. Εγώ θα ήθελα να πω σήμερα, όπως λέμε σε κάποιο φίλο που κάνει κάποιο σάλμα, σταμάτα, σταμάτα μην κάνεις αυτή τη μεγάλη βλαγία. Ίσως σήμερα οι δήμαρχοι που πραγματικά είναι πραγματιστές, έχουν τα πόδια που πατάνε στερεά στο έδαφος και βλέπουν την κατάσταση, πρέπει να ενεργήσουν διαφορετικά. ένα συνάδελφος ότι έγιναν χειραγωγήσεις από εξωτερικές δυνάμεις. Δεν το διαπίστωσαν οι Βρετανοί, άρα μπορούν να οπισθοδρομήσουν πριν από τις 29 Μαρτίου να κάνουν ένα νέο δημοψήφισμα ώστε να αποφευθεί το Brexit, το οποίο θα έχει μόνο αρνητικές ε, επιπτώσεις και θα κατακαιρματίσει την Ευρώπη. Θα είναι καταστροφικό για τη Μεγάλη Βρετανία. Και μετά από την ε, ε, Μεγάλη Βρετανία, εάν χάσει, χαθεί και η Ουαλία ή η Σκοτία, θα γίνει μια μικρή περιφέρεια μέσα στη χώρα του η Μεγάλη Βρετανία. Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε τόσο έντονα συγκινησιακό περιβάλλον. Είναι η τελευταία συνεδρίασή μας πριν από την 29η Μαρτίου. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να καταλήξω σε, το, σε, ε, σε συμπεράσματα, διότι υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες. Ούτως ή άλλως το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε και στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής, της Επιτροπής μας τον Απρίλιο και στην τελευταία μας συνάντηση. Είμαστε όμως όλοι πεπισμένοι ότι πρέπει και θα βρούμε την ε, κατάλληλη φόρμουλα για να συνεχίσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία με τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχάς είχαμε προβλέψει συζήτηση για την Επιτροπή Γειτονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυρία Μογκερίνη. Δυστυχώς όμως μετά από την πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα χρειάστηκε να πάει στην συνεδρίαση της ομάδας επαφής στο Μοντεβίδεο. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να κάνουμε συζήτηση για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο Φρανσουά Αλμπέχα Μισιά, πρόεδρο του Συμβουλίου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων τη Δυτικοφραϊκής Οικονομικής και Νομισματική Ένωση και υπουργό τη χώρα, το οποίο ε, ήταν στην συνάντηση που οργανώσαμε αυτή την εβδομάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον οποίο ε, καλωσορίζω θερμά σήμερα εδώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνετε πόσο μας καίει το θέμα του Brexit έγιναν στη συνάντηση που κάναμε περίπου 660 άτομα που εκπροσωπούν την ε, ε, ε αποκεντρωμένη τοπική και ε, περιφερειακή διοίκηση. Όλα αυτά έγιναν για να μπορέσουν να γίνουν συζητήσεις για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην μεγάλη πρόκληση στα πλαίσια της αηφόρου ανάπτυξης και βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη τι προβλέπει ο προπολογισμό του 2020. Τα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας πρέπει να είμαστε ενεργοί και μέσω εταιρικών σχέσεων να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που τίθενται στον πλανήτη μας διότι καθορίζουν την ε, αηφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και παρεθνικό επίπεδο. Οι περισσότεροι στόχοι της εφόρου ανάπτυξης εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την βούληση και την δυνατότητα των περιοχών να μπορέσουν σε επικεντρωμένο επίπεδο να αποτυπωκριθούν σε κάτι τέτοιο. Η σημασία τους θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να αντικατοπτρίζεται στα πλαίσια της σφαιρικής γενικής πολιτικής και στα πλαίσια της υποστήριξης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το ψήφισμα του συναδέλφου μας το σχετικό του κ. Γιάσεν το Δεκέμβριο έριξε Ποιο είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και πρέπει να πω ότι έγινε θετικά αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο συμπεριέλευε στο σχέδιο έκθεση που έκανε σχετικά με το θέμα αυτό. Τελικά η υποστήριξη στην αποκεντρωμένη συνεργασία περνάει και από την ε, συνεργασία που θα κάνουμε και πάλι στα πλαίσια της σχέσης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους μέσω σφιγμομετρήσεων απόψεων ε, στις οποίες θα ήθελα να συμμετάσχετε ενεργά θα δούμε και ποιες είναι οι δικές σας απόψεις και μπορείτε αυτό να το κάνετε με τη συνδρομή της γραμματείας έξω από την αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο ε, Υπουργό κύριο Αμισά Αλμπέρ, που είναι και πρόεδρο του Συμβουλίου Τοπικών Αυτοδικήσεων Δικοτικοφρικής Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στα πλαίσια τη συνεργασία που έχουμε, κύριε ε, Υπουργέ, θα μα πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το φόρουμ και μετά από εσά θα δώσω το λόγο σε άλλα μέλη του φόρουμ και όσους συναδέλφους έχουν εγγραφεί για την ε, θέμα αυτό. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής Περιφερειών, κυρίες και κύριοι, ηγήθηκα της αντιπροσωπείας των τοπικών αυτοδιοίκησεων Ινδικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση και σα πω ότι χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σα για να μπορέσω να ανταλλάξω απόψη για ένα θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Δηλαδή την συνεισφορά των πόλεων και των περιφερειών στην ανάπτυξη. Δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα αυτό χωρίς να σας μιλήσω για τα διδάγματα του φόρουμ πόλεις και περιφέρειες για την συνεργασία για την ανάπτυξη που έλαβε χώρα τη Θέρκη την Τρίτη στις Βρυξέλλες. Το φόρουμ αυτό είναι ένας χώρος διαλόγου μοναδικός για την ε, ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι των ε, τοπικών και περιφερειακών αργών της Ευρωπαϊκής και των χωρών που, των χωρών που συμμετέχουν ως εταίροι καθώς και δίκτυα πόλεων, ενώσεις, που ενδιαφέρονται για το όλο θέμα συζήτησαν αυτό το τόσο σημαντική σημασία ε, ε, θέμα που είναι η αηφόρος αστική ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικό περιβάλλον εφεξής ενώ το 1960 περίπου το 34%. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τρόπο εξαιρετικό. Το θέμα αυτό το συζήτησαν οι διάφοροι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Open Space. 60 περίπου διαφορετικά θέματα συζητήθηκαν ε, από την ε, αλληλέγγυο οικονομία μέχρι την συμπεριληπτική διακυβέρνηση. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους συμμετέχοντες που έκαναν ό,τι μπορούσαν στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων για την ποιότητα των συστάσεων που έστειλαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης, ε, πρέπει να πω ότι κατά πρώτο λόγο οι εκπρόσωποι συνέστηναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προσέχει με ε, ιδιαίτερα την ε, διαφορετικό, το διαφορετικό χαρακτήρα και την ποικιλία των διαφόρων επικρατειών που καλύπτονται από την δική της αναπτυξιακή πολιτική. Πρέπει να πω ότι κάθε χώρα έχει τις ε, ιδιαιτερότητές της. Στον Ήγηρα, Φερρυπίν, ένα από τα ε, συστατικά κράτη της ε, Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Έχουμε το 83,63 των ατόμων που ζούσαν το 2017 που έγινε μετρήσεις σε υπαίθριε περιοχές. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια των διαφορετικών χαρακτηριστικών που έχει κάθε περιοχή. Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι κατάλληλες ανεπτυξιακές πολιτικές και όπως ε, θα αναφέρω σε ένα παράδειγμα με μικρά σχέδια με λίγους ε, χρηματικούς πόρους που δίθενται, που διατίθενται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει κάποια, ε, κάθε μικρή τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, παράδειγμα η μικρή πόλη του Ντόγκμπο στο Μπενέν και η βέλγικη πόλη του Ροζλάρ που είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα αποτελεσματικού προγραμματισμού παρά το περιορισμένο ε, περιορισμένα κονδύλια που είχαν, δηλαδή για πέντε χρόνια 120.000 ευρώ. Πάρα πολλοί ε, συμμετέχοντες μίλησαν για το θέμα της χρηματοδότησης της αποκεντρωμένης συνεργασίας. Και πρέπει να πω ότι πρέπει να δούμε του καθενός τις ε, ε, ιδιαιτερότητες και πάλι. Ποιες ήταν οι διάφορες συστάσεις που έγιναν. Η αηφόρος αστική ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη σημαντικά στοιχεία όπως την απασχόληση, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ενσωμάτωση των μεταναστών και άλλα θέματα. Θα αναφέρω τα πιο σημαντικά. Πολλοί μίλησαν για την ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε κυρίως στους νέους. Δεύτερον, ο ρόλος των γυναικών που είναι υπέρ της ανάπτυξης. Πολλές φορές αναφέρθηκε το θέμα αυτό και πρέπει να πω ότι η σύσταση είναι να υποστηριχθούν τα δίκτυα των γυναικών για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν ακόμη περισσότερο στις αγορές εργασίας η πρόσβασή τους σε θέσεις ευθύνης και βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών που ε, αφορούν κυρίως τις γυναίκες. Κατά τρίτον, δεν μπορώ να μην αναφέρω και το θέμα των εκριζωμένων λαών. Από τις διάφορες ανταλλαγές απόψεις που έγιναν και από την λογική εταιρική σχέση στα πλαίσια της αποκεντρωμένης συνεργασίας δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για την στρατηγική σημασίας ανάγκη να αλλάξουμε όλη την έννοια και την αντίληψη ε, που αφορά την μετανάστευση κρίσης, να την κάνουμε μετανάστευση για να ανοίξουν νέες δυνατότητες. Κυρίες και κύριοι, είμαι πεπισμένος ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για προκλήσεις σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορέσουν να σας είναι χρήσιμες. Ελπίζω ότι οι συστάσεις οι οποίες υπευλήθηκαν από τους συμμετέχουν θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν την εργασία την οποία επιτελούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω όλους ιδιαίτερου από τα μέλη τη Επιτροπής Περιφερειών να μην αφήσουν τις συστάσεις της κοινότητα για την συνεργασία και την ανάπτυξη να παραμείνουν θεωρητικά σε ένα σιρτάρι Άρα να τους θέσουν σε πράξη και να εντάξουν στα πλαίσια του δυνατού στις ε, νομοθετικό έργο το οποίο επιτελείται στις Βρυξέλλες ώστε να μπορέσουν στην περιοχή του καθενός να αποτελέσουν συγκεκριμένη ε, δημόσια πολιτική υπέρ της ανάπτυξης των λαών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτή την ε, προοπτική την οποία σκιαγραφίσατε, για τα συμπεράσματα που μας παρουσιάσατε και αρχίζει η συζήτηση ο συνάδελφος Βιτσέντσο Μπιάνκο είναι από εμάς ο πρώτος συνάδελφος που θα λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μίχα, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας η οποία επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο τον ΟΤΑ σε όλη του την ποικιλομορφία για να ανταποκριθούν ακριβώς την τοπική ανάπτυξη και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Έχουμε λοιπόν το Φόρουμ ε, Πόλεων και Δήμων ε, για την Ανάπτυξη που οργανώσαμε Δευτέρα και Τρίτη με την Κομισιόν και εκεί πέρα είχαμε γύρω στους 500 συμμετέχοντες από 80 σχεδόν χώρες από τις 5 υπήρους. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει η Επιτροπή μας σε αυτό το θέμα. Είχαμε λοιπόν εκπροσώπου από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων 50 μέλη τη Επιτροπή μα, αλλά και τον δήμαρχο του Μογκαντήσου, τον δήμαρχο ε, του Ισλαμαμπάντα, της Εμπνομπένχα, ε, τη ε, Τίνιδας ή δήμαρχος μάλιστα είναι γυναίκα για πρώτη φορά ε, επιφανείς εκπρόσωποι επίσης ε, του επιστημονικού κόσμου το φόρουμ μας ε, προσέφερε πολλές δυνατότητες ακριβώς για διμερείς επαφές. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση σε έναν ανοιχτό χώρο και ζητήσαμε να υπάρχει μια ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών ε, και σκέψεων σε 60 ομάδες ε, εργασίας να ανταλλάξουμε εμπειρίες ε, όσον αφορά την αποκεντρωμένη συνεργασία και βεβαίω να γίνουν πολιτικές συστάσεις απευθυνόμενε σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωση ω μια άμεση απάντηση σε αυτή τη σύσταση η Κομισιόν έλαβε υπόψη την εταιρική αυτή σχέση. Συμπερασματικά, Πρόεδρε, η άγνοια και οι προκαταλήψει ε, συχνά ε, πακιδεύουν τον φόβο, το, ε, την στάση με... μάλλον δεν βοηθούν στο να υπάρχει μια ελπίδα στο να κοιτούμε προς το μέλλον με θετικό τρόπο και ε, είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για προβλήματα που είναι πολύ πιο κοινά και πολύ πιο συνηθισμένα από αυτό που θεωρούμε ή πιστεύουμε. Σας ευχαριστώ ο κύριος ε, Λόπες Μοίρας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε αμυσιά. Νομίζω ότι ως πολιτική υπεύθυνη και προκειμένου να προωθήσουμε το κοινά συμπεφωνημένο θεματολόγιο δεν μπορούμε να δράσουμε μεμονωμένα, απομονωμένα ο ένας φορέας από τον άλλον. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε γνώσεις, τεχνολογία, βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να προωθήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδιαίτερα στην, ε, στο νότο, στην Μεσογειακή, στο μεσογειακό τμήμα της Ευρώπης, των περιφερειών μας, έχουμε στην ε, Μεσόγειο, έχουμε στη Μούρθια από την οποία προέρχομαι, ε, συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε με, με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους υδάτινους πόρους μας, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η συνεργασία λοιπόν η διαπεριφερειακή με πολύ σημαντικά έργα που εξασφαλίζουν την ε, βιώσιμη ε, καλλιέργεια και γεωργία στο νότο της Ευρώπης θα πρέπει να μπορέσουμε να προσφέρουμε μέσα που θα εξασφαλίζουν την επιστηστική ασφάλεια και την συνέχιση της βιώσιμης καλλιέργειας μας. Νομίζω ότι έχουμε ε, την ευκαιρία σήμερα με την παρουσία του κυρίου Αμισιά ε, για μια καλύτερη συνεργασία και ανάπτυξη με τους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή των Περιφερειών, των περιφερειών και προς τους οποίους έχει δεσμευθεί η περιφερεια της Μούρθια. Επομένως, μέσω της υλοποίησης κοινών συμπεφωνημένα ε, συμπεφωνημένα ε, ε, κατευθύνσεων μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο πρόεδρος. Τον λόγο έχει ο κύριος Σίμονς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η κυρία Μπέντλεϊ νομίζω ότι πολύ καλά περιέγραψε την προετοιμασία που κάνουμε για το Brexit και η προσέγγιση είναι πώς μπορούμε να εστιαστούμε σε εκείνα τα στοιχεία που θα έχουν τον ε, πιο θετικό αντίκτυπο στους πολίτες. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσει κανείς. Εγώ είχα την ε, ευκαιρία να επισκεφθώ ε, την ακτή ελεφαντοστού πέρυσι και είδα κάποιες από τις ωφέλειες του ευρωπαϊκού έργου και της ευρωπαϊκής βοήθειας προς τη χώρα αυτή. Νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινά εποφελές πλαίσιο για αναπτυξιακές ευκαιρίες. Έχουμε γεωργικά προϊόντα για τα οποία υπάρχει σημαντική ζήτηση εδώ στην Ευρώπη, στη χώρα αυτή και στις περιφέρειες εκείνες. Οργανική καλλιέργεια σοκολάτας και καφέ, για παράδειγμα, που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στην ακτή ελεφαντοστού και εποφελεί ε, σχέσεις ε, επιχειρήσεων εδώ στην Ευρώπη. Άλλη μια διάσταση που είναι σημαντική του έργου αυτού είναι κάτι που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στην αίθουσα. Πώς δηλαδή αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των παραγόντων που συνεισφέρουν στην ε, μαζική μετανάστευση. Η οικονομική ανάπτυξη δίνει τις ευκαιρίες στους πολίτες των χωρών αυτών και είναι ένας ο πιο σημαντικός ίσως παράγοντας. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά και θέλω να πιστεύω ότι κοιτώντα προς το μέλλον και πέραν συμφωνία τη Κοτονού, ότι θα εστιαστούμε στο πώς η δική μας προσέγγιση με την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου εντός ή εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι να αναπτύξουμε αμοιβαία εποφελείς εμπορικές σχέσεις και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούρτς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, θεωρώ ότι στην Ευρώπη, πέρα από τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο λέγεται η ανάπτυξη της Αφρικής. Είναι υπαρξιακή σημασία για την Ευρώπη. Η UNCTAD του ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι ανάγκες μέχρι το 2030 είναι 1,33 εκατομμύρια επενδύσεις για ανάπτυξη στην Αφρική. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Δηλαδή απαιτείται επιγόντως ο ιδιωτικός τομέας ε, να αναπτύξει μια στρατηγική η οποία θα είναι αποτελεσματική για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Δήμους ε, στην αναπτυξιακή εργασία. Ο Νικέα αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των Δήμων που διακρίνονται από τους άλλους φορείς ε, έχουν ε, και συγκεκριμένη πείρα για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα επί τόπου ε, και βεβαίω μπορούν να την μεταφέρουν υπάρχει και η άμεση επαφή με τον πολίτη μπορούν παραδείγματος χάρη να περιληφθούν και οι τοπικές ε, κοινότητες μεταναστών ε, και να δούμε μια διαφορετική επίδραση. Έτσι λοιπόν η συμπερίληψη των Δήμων είναι ένα μέσο για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή των Περιφερειών να δώσει εδώ πέρα κάποιες οθήσεις, ε, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερος επενεταίο. Και βεβαίω όλα αυτά δεν μπορούν παρά να είναι μια πρώτη προσέγγιση σε μια σαφώς πιο ισχυρή χρηματοδότηση στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Φραντ Σάουνσμπέργκερ τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αμίκια, ως εκπρόσωπος ε, μιας ε, ε, περιφέρειας στην κεντρική Ευρώπη θα ήθελα να πω πως δεν είναι μόνο οι χώρες της Μεσογείου οι οποίες έχουν κάποιες ευθύνες αλλά βεβαίως λόγω και των ιστορικών εξελίξεων ολόκληρη η Ευρώπη έχει ευθύνη απέναντι στην Αφρική. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει ακριβώς η, η Αφρική να αναλάβει το μέλλον ε, στα χέρια της ευτυχώς. Σημαντικό όμως ε, για εμάς είναι για τους ΟΤΑ το ότι έχουμε ένα συμβούλιο των τοπικών αρχών και έχει κάποιες ε, λειτουργίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να προωθεί και τους κοινωνικούς στόχους ε, της θέσης εργασίας, την εκπαίδευση βεβαίως, την εμβάθυνση της δημοκρατίας Η αναπτυξιακή πολιτική, κυρίες ε, και κύριοι, δεν είναι μόνο ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και των περιφερειών και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να υπάρξει άμεση βοήθεια από τις περιφέρειες της Ευρώπης στην Αφρική για να πάει η βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται στους Δήμους και τις περιφέρειες κυρίως αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Αμίκια, τα προβλήματα αυτά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, και να αντιμετωπίσουμε έτσι τις αιτίες της μετανάστευσης. Επίσης, η Αυστριακή Προεδρία τον Δεκέμβριο, όπως ξέρετε, οργάνωσε μια σύνοδο κορυφής ε, με την Αφρική για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες επενδύσεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Ελόνσα Σουμπήρια. Αγαπητέ Υπουργέ, έχουμε μια επίγουσα ανάγκη να καταπολεμήσουμε την ένδια η βασκική τοπική κυβέρνηση ε, πιστεύει ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την πραγματικότητα και όπως το κάνουμε εδώ και τρεις δεκαετίες μπορούμε πιστεύουμε να αναπτύξουμε αναπτυξιακές πολιτικές που να έχουν αυτά αποτελέσματα. Τον περασμένο έτος ε, ενίσχυσε με 48 εκατομμύρια διάφορες χώρες του Νότου η τοπική βασική κυβέρνηση χρηματοδοτώντας και πολλά ανθρωπιστικά έργα. Η συνεργασία μας η αναπτυξιακή ακολουθεί την αποκεντρωμένη κατεύθυνση του, του σχεδιασμού των πολιτικών μας. Βοηθάει κοινωνίες να διασυνδέονται και προωθεί έργα συνεργασίες μεταξύ των βασικών και των τοπικών φορέων. Και όλα αυτά περνούν από την κοινωνία των πολιτών στη χώρα των Βάσκων, που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση και εφαρμογή των έργων αυτών. Επίσης δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ισότητα των φύλων, στην βιωσιμότητα την οικολογική, στην ε, υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμής η κύρια εστίασή μας υπήρξε η Νότια Αμερική. Μόλις εγκρίναμε την ε, ε, τον πραγματισμό της περίοδου 18-22 που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις ε, στο επίπεδο της συνέπειας ε, της πολιτικής και στην συνέχιση της βοήθειας προς την Αφρικανική Ήπειρο. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε να το κάνουμε με διάφορες χώρες και της Νοτιοαμερικής και της Αφρικής στα πλαίσια της αναπτυξιακής αυτής πολιτικής. Μάλιστα, το λόγο έχει ο κύριος Άντλες Γιάντλα, που είναι ο τελευταίος ομιλητής σε αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχουμε το σύμφωνο των δημάρχων το οποίο έγινε παγκόσμιο και βεβαίω έχουμε δημιουργήσει και τον πρέσβη, τον θεσμό αυτόν και μια πολύ σημαντική συνεργασία με τις αφρικανικές πόλεις. Είχα βρεθεί προσφάτως στην Κένια και είδαμε κάποια πρόοδο στον τομέα της συνεργασίας και το ενδιαφέρον από την αφρικανική πλευρά είναι πάρα πολύ μεγάλο οι συνάδελφοι από τις ευρωπαϊκές πόλεις, ε, τις ε, περιφέρειες ε, μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα μαζί μας μέσω του συμφώνου των δημάρχων μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε και βεβαίως Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον τομέα της ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα καλέσω τον ε, κύριο Υπουργό τώρα να απαντήσει εφόσον το επιθυμεί. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους παριστάμενους και φυσικά όσους όλους παρενέβησαν σήμερα. Μας εξασφαλίζουν οι τοποθετήσεις σας για την βούληση της Επιτροπής των Περιφερειών να συνεχίσει την συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αφρικανικών χωρών. Πολλά έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πεδίο αυτό από πολλούς συλλογικού φορείς και μας είπατε σήμερα ότι θα εξακολουθήσετε να δημιουργείτε πλαίσια εταιρική συνεργασίας και είναι αυτό που επιθυμούμε και έχουμε ανάγκη. Ο κόσμος σήμερα δεν είναι απλώς πέντε ήπειροι, είναι ένα σύνολο ένα, μια συλλογική οντότητα ανθρώπων που ζουν στο έδαφος, σε αστικά κέντρα, στην, στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια και όπως είπε ένας από τους ομιλητές πρέπει να μάθουμε ένα τον άλλον για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα και νομίζω ότι η συμφωνία που υπεγράφει εδώ και μερικά χρόνια μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της κοινότητας Ουμόγια είναι ένα χρυσό παράδειγμα αποκεντρωμένης συνεργασίας και εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι οι τοπικοί φορείς ε, κάθε χρόνο που πηγαίνουν ε, και επισκέπτονται τις χώρες της Αφρικής για να σημειώσουν τι έχει υλοποιηθεί, τι έχουμε επιτύχει, πού υπάρχουν κενά, πού μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή αυτή. Όλες αυτές οι προσπάθειες δεν γίνονται απλώς για να αναπτύξουμε καλύτερα το πεδίο, το έδαφος, τον αστικό χώρο, αλλά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, των κατοίκων. Και έχουμε αντικείμενα θέματα ύψης της σημασίας, όπως η απασχόληση και κυρίως η απασχόληση των νέων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την Αφρικανική Ήπειρο για να έρθουν στην Ευρώπη είναι ανθρώπινοι πόροι που χάνει η Αφρικανική Ήπειρος. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση όχι στις χώρες αλλά στους πολίτες των χωρών αυτών ώστε να αναπτύξουν καλύτερα την δική τους οικονομία, τη δική τους ζωή και είναι οι τοπικοί φορείς εκείνοι που είναι οι πιο κοντινοί στους πολίτες και που μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Εάν στοχεύσουμε καλύτερα την βοήθεια αυτή, την ενίσχυση αυτή, γιατί πάνω από το ίμιση του συνολικού αφρικανικού πληθυσμού είναι νεαροί άντρες και γυναίκες, θα έχουμε πετύχει σε, μεγάλη, σε μεγάλο ποσοστό τους στόχους που έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Και πρέπει να δημιουργήσουμε και τις καλύτερες συνθήκες για να υποδεχθούμε καλύτερα τους ανθρώπους που μετακινούνται από την μία χώρα στην άλλη. Πρόκειται για φαινόμενα παλαιότατα και τα γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο σήμερα. Η κοινή μας παράδοση, η κοινή μας ιστορία μπορεί να μας βοηθήσει για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε το πρόβλημα αυτό της μετανάστευσης να μην είναι πρόβλημα πλέον, να πάψει να είναι πρόβλημα, αλλά να είναι ένα θετικό στοιχείο συνεργασία μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Ο κ. Λόπες αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο των αστικών κέντρων. Είναι προφανέ και είναι ουσιαστικότατη σημασία. Ο κ. Ντέιβιτ Σίμονς είπε πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να είναι υποφελέ για του πολίτε. Ε, χαίρομαι για την συνεχιζόμενη προσπάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αφρική. Ο κύριος Κούρτς, ο κύριος Γιάντλερ και άλλοι ομιλητές όλοι είπαν ότι θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή και την ενισχύσουν. Αυτό επιθυμούμε και εμείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και να εκφράσω την ελπίδα ότι η αποκεντρωμένη αυτή συνεργασία θα μπορέσει να φτάσει στην πλειοψηφία ένθεν κακήθεν των υπήρων μας, ώστε αυτές οι γέφυρες που θέλουμε να οικοδομήσουμε μεταξύ Βορρά και Νότου να μην είναι μόνο μεταξύ κρατών, γιατί όπως είπαν και αρκετοί ομιλητές, η πραγματική συνεργασία διεξάγεται πιο αποτελεσματικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και επομένως ο ρόλος σας ημών με ύψιλον του Βορρά και ημών με ήττα του Νότου είναι να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε οι μελλοντικέ γενναίε, τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζουν σε έναν κόσμο αλληλέγγυο, δίκαιο και ασφαλή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ, για την ε, ενεργό σας ε, συμμετοχή στη συζήτηση. Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω κατά 200% τα όσα είπατε. Είμαι σίγουρος και ότι θα συνεχίσουμε την αποτελεσματική μας συνεργασία με τρόπο βιώσιμο. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε ακόμα τρει νομοδοτήσεις προς έγκριση και πάμε αμέσω στο 8ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον με εισηγητή τον κύριο Λάμερς, τον οποίον καλό να προσέλθει στο βήμα.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 Avant Πρωτού δώσω το λόγο στον εισηγητή μα. να καλωσορίσω την, ε, το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βαλεάν που θα συμμετάσχει στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Βουλευτή. Monsieur ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την συνάδελφο εδώ πέρα, την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που βρίσκεται εδώ πέρα στην παρουσίαση αυτής της έκθεσης βρισκόμαστε στην προκαταρκτική φάση της ε, νέας ε, πολιτικής ε, κλίματος και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το πρώτο θεσμικό όργανο το οποίο εκφράζεται Ήδη έχει υπάρξει αξιολόγηση του εβδόμου του προηγούμενου προγράμματος ε, δράσης ε, από το Κοινοβουλίο. Η Κομισιόν ακόμα δεν την έχει ετοιμάσει, όμως ε, έχουμε μια μεγάλη παράδοση στην σύνταξη γνώμοδοτήσεων για το κλίμα και το περιβάλλον στα λεγόμενα αυτά σχέδια δράσης για το περιβάλλον και το έβδομο πρόγραμμα το οποίο αξιολογείται αποτελεί για μένα την βάση για να κοιτάξουμε στην ε, επόμενη φάση. Διαπιστώνουμε λοιπόν μετά από 40 χρόνια ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον πως έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. Ε, είναι διαφορετικό πράγμα οι κανόνες από την εφαρμογή και δυστυχώς δεν βλέπουμε πάντα τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Μπορούμε μάλιστα να μιλάμε για ένα κενό εφαρμογής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της κατάρτισης σχεδίων και κανόνων και από την άλλη πλευρά των δράσεων για να μπορέσουμε ακριβώς να δούμε την αηφορία της παραγωγής και της κατανάλωσης. Δεν μπορούμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό να το λύσουμε με τις νοοτροπίες του χτες θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και ένα διαφορετικό σύστημα, κάτι το οποίο είναι επίσης μια μετάβαση. Η πρότασή μου λοιπόν περιέχει κάποιες ε, τέτοιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φύγουμε από την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αντιμετώπιση των αιτιών. Και αυτό πάντα σε συνεργασία με την βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα. Κατόπιν θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με την μετάβαση της οικονομίας, ε, της ενέργειας, της κινητικότητας ε, των τροφίμων. Είναι μεγάλες υποθέσεις ε, αυτές και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν με τους παραδοσιακούς τρόπους και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη χρηματοδότηση από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή και μια ολιστική αντιμετώπιση. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως ε, τα προβλήματα αυτά όσον αφορά την συνοχή της πολιτικής είναι ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος συχνά αντιμετωπίζουν ε, και έχουν να ανταγωνιστούν τα οικονομικά ζητήματα. Να Έχουμε από την άλλη πλευρά λοιπόν την προσέγγιση της υγιεινής ζωής και μιλάμε για την υγεία και του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και της φύσης και να μην τα βλέπουμε ως ξεχωριστούς πυλώνες ε, μονοδιάστατης πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ιδιαίτερος η εθνική προσέγγιση για τις πόλεις ε, και χωριά και τις περιφέρειες που παίζουν σημαντικό ρόλο και η ΟΤΑ ακριβώς ε, είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι κινούνται και εργάζονται και έχουν ε, και μεγάλη σημασία αλλά αποτελούν και μεγάλο, κόσμο, μεγάλο τμήμα της ρήπανση η οποία παράγεται η μετάβαση στον τομέα των μεταφορών αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση ειδικά για την ε, Ήπεθρο θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες λύσεις και κάθε περιφέρεια θα πρέπει να είναι φιλόδοξη για να κάνει αυτό το οποίο είναι σε θέση να κάνει καλύτερα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους αδέλφους που υπέβαλαν ε, τροπολογίες τις οποίες ε, προσπάθησα να ενσωματώσω στις δικές μου τροπολογίες για να είναι κάπως πιο ωραίο το κείμενο και βεβαίω αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης και για μένα ένα σημαντικός ε, πυλώνας, μια χρήσιμη μέθοδος για μια πιο ολιστική άσκηση πολιτικής. Ε, αλλά δεν είναι δυνατόν να μπει σε όλες τις παραγράφους αυτής της έκθεσης. Ε, το δέχτηκα σε κάποιες ε, τροπολογίες όπου έχει κρίσιμο ρόλο και νομίζω έχουμε μια καλή αφετηρία και σας ευχαριστώ για την στήριξή σας επίσης. κάποιες από τις ε, τροπολογίες αυτές. Ε, δεν την δέχτηκα γιατί δεν έχουν τελικά θέση σε αυτήν την ε, έκθεση. Αλλά μου είπαν οι συνάδελφοι ότι μπορούν να συμβιβαστούν με τις τροπολογίες οποίες πρότεινα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την στήριξη που μου έδωσε για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις ε, στο τοπικό επίπεδο με υγιείς ανθρώπους, ε, υγιές περιβάλλον, υγιή οικονομία τελικά και ζωή για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Συγητή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ευρωβουλευτή επικεφαλής της ε, Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και Ασφαλείας Τροφίμων, την κυρία Βαλεάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω ε, εσάς, κύριε Καλχάιντς Λάμπερτς, για την ευγενική σας πρόσκληση και τον κύριο Λάμερς, τον εισηγητή, για την μελέτη του στα πλαίσια του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτική και το σχέδιο δράσης μπορούν μόνο ε, να υλοποιηθούν αποτελεσματικά σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο. Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένας ζωτικός κόμβος σε αυτήν την προσπάθεια υλοποίησης. Αν δείτε ουσιαστικά τμήματα του, του προγράμματος, καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, καλύτερη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους φορείς, ε, βιωσιμότητα ενισχυμένη για τα στατικά κέντρα, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε τη μέγιστη συμμετοχικότητα των Δήμων και Περιφερειών προκειμένου να εφαρμόσουμε τις περιβαλλοντικές μας πολιτικές. Επομένως με χαρά σήμερα συμμετέχω σε αυτήν την επίκαιρη συνάντηση που έχετε για να συζητήσουμε το πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2020. Μερικοί σχολιαστές επικρίνουν την ευρωπαϊκή πολιτική γιατί μερικές φορές ε, ε, φαίνεται να έχει ιδιαίτερα γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Και ίσως ε, κάποιοι δήμοι δίνουν την εντύπωση ότι στέκονται στην πρόοδο των πολιτικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια αξιόπιστη ανάλυση, μελέτη του τι πρέπει να αλλάξει και τι όχι. Προτού δούμε λοιπόν το μέλλον του περιβαλλοντικού προγράμματος, του πρόγραμματος δράσης, θα ήθελα ε, να δούμε λιγάκι τα διδάγματα από το υφιστάμενο πρόγραμμα. Θα βασίσω το σχόλιά μου ε, στη βάση του γεγονότος ότι η Επιτροπή ΕΝΒΗ προχώρησε στη δική της ενδιάμεση ε, αναθεώρηση της υλοποίησης του προγράμματος για να εντοπίσει τις ελλείψεις, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την κατεύθυνση, την πορεία του, για να δούμε τι καλύτερα πρέπει να κάνουμε στον επόμενο προγραμματισμό. Τα βασικότερα πορίσματα της αξιολόγησής μας, της εξέτασης αυτής, ήταν διάφορα μέσα πολιτικής υπό το πρόγραμμα αυτό, ότι είναι περιορισμένης έκτασης και επομένως τα αποτελέσματα είναι σε μια σειρά περιοχών μη ικανοποιητικά. Οι περιοχέ που φαίνονται πιο προβληματικές ως προς την υλοποίηση είναι το πεδίο τη βιοπικιλότητα, διαχείρισης των απορριμμάτων, η ποιότητα του αέρα και η χορύπανση. Η χρηματοδότηση φαίνεται να είναι ανεπαρκής ως προς τις πραγματικές ανάγκες. Θα τα δούμε ένα προς ένα. Για την βιοπικιλότητα θεωρώ ότι η συρρήκνωση Τη βιοπικιλότητας είναι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας. Δεδομένης της αξίας της για το οικοσύστημα και για την ανθρώπινη τελικώ υγεία και ευζοία, η προστασία της βιοπικιλότητας θα πρέπει να λάβει την περισσότερη πολιτική προσοχή που μπορούμε να δώσουμε. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος στην βιοποικιλότητα. Η ανακοίνωση της Κομισιόν για την στρατηγική βιοποικιλότητας είναι καλοδεχούμενη προκειμένου να καλύψουμε τα κενά μας, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τις ίδιες ε, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην ποιότητα του αέρα, είναι προφανές ότι η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι όσο πιο καθαρή γίνεται, ο αέρας που αναπνέουμε δηλαδή, και συχνά οι τοπικές ε, αρχές, οι τοπικοί φορείς αναγκάζονται να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Να θυμίσω ότι τα θύματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι περισσότερα από τα θύματα στα οδικά ατυχήματα. Έχουμε άνω των 400.000 πρώιμους θανάτους το έτος. Επομένως είναι επίγουσα η ανάγκη της βελτίωσης της ε, ατμοσφαιρικής ποιότητας στην Ευρώπη, της ποιότητας του αέρα, που συμφώνησαν τα κρατημέλη και το Κοινοβούλιο ήδη προδεκαετίας. Άλλη μια περιοχή όπου μπορούμε σημαντικά να βελτιωθούμε είναι η συνέπεια προς άλλα προγράμματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο ότι αυτού του είδους τα σχέδια δράσης θα υλοποιούνται αποτελεσματικά, αλλά ότι θα είναι συνεπή και προσαρμοσμένα με, την, ε, με το μακρόπνο όραμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Θεματολόγιο 2030, τους στόχους βιωσιμού ανάπτυξης και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί σε συνέδρια όπως η ΚΟΠΣ και άλλα διεθνή φόρα. Ένα πεδίο που είναι κλειδί είναι ο τομέας των μεταφορών. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα εξακολουθούν να αυξάνονται και εντός ενός έτους μεταξύ του 17 και του 18 η Κομισιόν εξέδωσε άνω των 12 νομοθετικές προτάσεις για τον ε, τομέα των μεταφορών προκειμένου να κινηθούμε σε καθαρές μεταφορές μέχρι τα μέσα του αιώνα. Μεταξύ αυτών επιτύχαμε ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα με το 35,5% των εκπομπών διοξιδίου για νέα αυτοκίνητα και 31% για μικρά φορτηγά μέχρι το 2030 και είμαστε στο τελευταίο τμήμα των διαπραγματεύσεων για την μείωση των εκπομπών για τα φορτηγά. Έχουμε αυξήσει το, πεδίο, το επίπεδο της φιλοδοξίας μας και στους δύο φακέλους γιατί χρειαζόμαστε εύρος στους στόχους όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον πλανήτη αλλά για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Η τάση προς καθαρά οχήματα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν μπορεί ο δικός μας κλάδος να μείνει πίσω. Στα θετικά του ισολογισμού η μελέτη του Κοινοβουλίου σημειώνει ότι η πολιτική αυτή εξακολουθεί να είναι ένα πολύτιμο μέσο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλους τους μακροπρόθεσμους στόχους, τους περιβαλλοντικούς και στο κλίμα. Και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να διαθρώνονται σε βραχυπρόθεσμες απτές πολιτικές που θα μπορούν να υλοποιούνται και να ελέγχονται, να παρακολουθούνται αποτελεσματικά. Και θα ήθελα εδώ να στραφώ σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με το 8ο αυτό σχέδιο δράσης. Καταρχά πρέπει να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα στην, ε, την Κομισιόν. Μην καθυστερείτε ε, ε, στο 8ο σχέδιο δράσης. Πρόγραμμα δράσης. Η Κομισιόν μόλις τώρα ολοκληρώνει την τελική της αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν το Μάιο. Η προετοιμασία του 8ου προγράμματος θα πρέπει να είναι προχωρημένη γιατί χρειαζόμαστε ένα λειτουργικό έτοιμο πρόγραμμα από 1η Ιανουαρίου που θα πρέπει να είναι συνεπές προς άλλες πολιτικές. Η προσέγγιση σάιλο της Κομισιόν είναι ξεπερασμένη πλέον διότι θα πρέπει να συσχετίζεται με άλλε προτεραιότητες αποτελεσματικά και οργανικά το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, το μελλοντικό πρόγραμμα δεν θα πρέπει πρώτα να συνδέεται με άλλα έργα και προγράμματα, αλλά να θεμελιώνεται στους μακροπόθεσμους στόχους. Έχουμε μια δύσκολη συζήτηση μπροστά μας για την κατάλληλη κατεύθυνση ώστε να απομακρυνθεί η οικονομία από τον άνθρακα. Είχαμε και την ανακοίνωση πέρυσι της Κομισιόν για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική αυτή και ψήφισμα που θα έχουμε από το Κοινοβούλιο το Μάρτιο σχετικά με το θέμα. Ακριβώς προτού δηλαδή τεθεί το Κοινοβούλιο σε απόλυτη προεκλογική εκστρατεία. Αντίστοιχα θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν γιατί το εθνικό επίπεδο είναι το σημείο συμφόρησης σχετικά με την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Χρειαζόμαστε επίσης καλύτερη ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τις περιφέρειες και που θα πρέπει να υλοποιηθεί από τις περιφέρειες. Διότι βεβαίως το επίπεδο το τοπικό και το περιφερειακό δεν μπορεί να περιμένει το κεντρικό επίπεδο προκειμένου να ενεργοποιηθεί και επομένως προσβλέπουμε και υπολογίζουμε στη δική σας ενεργό συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα αρχίσουμε τώρα τη γενική συζήτηση για το νομοδότηση αυτή. Πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στην κυρία Όλικα Χίλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Έχουμε υποβάλει πολλές ε, τροπολογίες ε, για την αηφορία και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι η στρατηγική αυτή η στόχη της ανάπτυξης ε, είναι μια αρχή για να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως είπε ο κύριος Λαμή, είναι σημαντικό να τα συνδέσουμε αυτά, περιβάλλον, αηφορία και υπ' αυτήν την έννοια σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ρόμπι Μπίβερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Βαλεάν για την ε, παρουσία σας. Θεωρώ ότι υπογραμμίζει και την καλή συνεργασία που έχουμε με το Κοινοβούλιο ειδικά για θέματα περιβάλλοντος και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Λάμερς για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε εδώ. Σημαντική αυτή η γνωμοδότηση, ειδικά στο θέμα προστασίας της φύσης του περιβάλλοντος. Έχουμε συνεργαστεί στις σχετικές οδηγίες με το Κοινοβούλιο, στην COP24, και η συνεργασία για τους ε, στόχους αυτούς είναι πολύ επικοδομητική. Ε, η απώλεια της βιοπικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι θέματα οποία και στατιστικά αν δείτε είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους ε, πολίτες μας και πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι πολύ θετικό το ότι οι νέοι ήδη είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι για αυτά τα ε, ζητήματα και έχουμε πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι εμείς ειδικά ως τοπικές αρχές ε, έχουμε πολλές δυνατότητες να δραστηριοποιηθούμε είτε μιλάμε για την απώλεια της βιοπικιλότητας στη γεωργία την καταστροφή της γεωργίας τα ζανιοκτώνα και η ρήπανση όλα αυτά παίζουν ρόλο και τα ανέφερε η κυρία Βαλεάν έχουμε ρήπανση του νερού, του εδάφους, του αέρα και φωτορύπανση και η φωτορύπανση είναι ε, κάτι το οποίο εκδιώκει τα είδη οπότε σας ευχαριστούμε κυρία Βαλεάν για την παρουσία σας και την περαιτέρω καλή συνεργασία ελπίζω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάδελφο Σέρτελ ζητάει το λόγο, δίδω αμέσω. Τη συνάδελφο λοιπόν το λόγο. Arvoisa puheenjohtaja, minä tulen Suomesta, Espoosta. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Φιλανδέζα είμαι εγώ από το ΕΣΠΟ και είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ε, τώρα. Με όρισαν και μου ζήτησαν να παρουσιάσω μια σχετική έκθεση. Οι 17 αυτοί στόχοι πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το 2030 όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Ελπίζω λοιπόν ε, στο 8ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα να συνεργαστούμε όπως κάναμε και στο σύμφωνο των δημάρχων. Θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω όλες τις πόλεις ε, και τις περιφέρειες να εφαρμόσουν αυτούς τους σημαντικούς ε, στόχους. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα, πολύ σημαντικά εργαλεία όταν πολεμάμε την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συνεργαστούν τα διάφορα επίπεδα της διοίκησης ε, με τους πολίτες ε, και τις εταιρείε. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και για την πολύ καλή συζήτηση που έχουμε εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ε, ζητά για τη γενική συν... ζήτησε κανείς άλλο το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και στην πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να απαντήσουν. Κύριε Ισηγητά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα πράγματα έχω να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπαν τα μέλη. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ε, συνεργασία και στην Επιτροπή και για τις ε, θετικές αντιδράσεις τους ε, σήμερα στην τελική εκδοχή αυτής της να πω λίγο κάτι για αυτό το οποίο είπε η κυρία Βαλίαν. Ακριβώ ε, σταθήκατε στο θέμα στο οποίο κάνει συστάσεις ε, και η δική μου η έκθεση. Δηλαδή το γεγονός ότι τα θέματα αυτά της ε, νομοθεσίας δεν καθορίζονται πάντα στο τοπικό επίπεδο και βεβαίως ε, δεν να ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είναι η μεγαλύτερη επίδραση. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε η πολιτική να κατευθύνεται στο τοπικό επίπεδο. Το επίπεδο λοιπόν της ευρωπαϊκής νομοσίας δεν χρειάζεται να αλλάξει αυτό το οποίο λέμε ως κεκτημένο για μένα είναι το ελάχιστο το οποίο πρέπει να εγγυόμαστε σε όλους τους πολίτες αλλά οι πόλεις, οι περιφέρειες πρέπει να έχουν την ε, δυνατότητα να είναι πιο φιλόδοξες ε, και γι' αυτό εξεπλάγει ε, θετικά από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι που ακριβώς τονίζουν την σημασία αυτού του θέματος. Και έχουμε την αξιολόγηση του 7ου σχεδίου δράσης που Βεβαίω θα αναλάβει η καινούρια κομισιόν σε μερικούς ε, μήνες και το καινούριο κοινοβούλιο και πραγματικά ελπίζω συνάδελφοι να είναι ευχαριστημένοι από αυτήν την έκθεση για να ε, περάσει μια διαφορετική νοοτροπία και στα γραφεία της ε, Κομισιόν και μια διαφορετική οργάνωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχετε εσείς, ε, κύριε Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως είναι η τελευταία φορά που έχουμε επισήμω κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειών για την προερωτική τη ε, ε, προσέγγιση, τον εισηγητή, για την πολύ επικοδομητικό ρόλο και σχέση που έχει με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας παρακαλέσω και να διατηρήσει την προσέγγιση και για την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα θέματα είναι εξίσου σημαντικά και για σας και για μας. Εσείς λοιπόν, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να είστε όλοι ενωμένοι, να είμαστε όλοι ενωμένοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη για την περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη. Εύχομαι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα φτάνουμε στην συζήτηση για τις τροπολογίες. Αρχίζουμε με την τροπολογία 1 του εισηγητού που αντικαθιστά την 1, 2 και 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 5 του Ισούγητου. Αντικαθιστά την 5, 6 και 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 του εισηγητού. Προ την κατάσταση τη αρχική 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προτείνω ομαδική τροπολογία για τι 10 και 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 12 του εισηγητού. Σε την κατάσταση της αρχικής 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13 του εισηγητού. Αντικαθιστά την 13, 14 και 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 16. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 του εισηγητού που αντικαθιστά την 17, 18, 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 20 του εισηγητού. Αντικαθιστά την αρχική 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 που αντικαθιστά την 21, 22 και 23. 21 είναι του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προτείνω ομαδική ψηφοφορία για την 24 και 25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27. Απορρίπτεται αν κατάλαβα καλά λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θέλετε το λόγο? Έχετε το λόγο κύριε Ριβέρς. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω ότι τις δύο τροπολογίες στο σημείο 29 τις βλέπουμε στο πλαίσιο των ε, νησιών και έτσι μπορούμε να τις ε, στήριξουμε βεβαίως οπότε θα τις υπερψηφίσουμε υπέρ ωραία υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ συγγνώμη 30 λέει ο πρόεδρος συγγνώμη υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται 31 υπέρ κατά εγκρίνεται 32 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ Λίγη ψηφοφορία εγκρίθηκε η τροπολογία 33 του εισηγητού που αντικαθιστά την ε, αρχική 33 υπέρ κατά εγκρίνεται. 35 του εισηγητού. Πάω πολύ γρήγορα, λέει ο πρόεδρο. Ξέχασε την 34. Υπέρ τη 34, κατά. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στο 35 του εισηγητού που αντικαθιστά 35, 36 και 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά απορρίπτεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 του εισηγητού που αντικαθιστά την προηγούμενη υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται Η 43 του εισηγητή αντικαθιστά την αρχική 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ κατά απορρίπτεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ τη γνωμοδότηση. Κατά. ποιο απέχει. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά για την εργασία σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάνουμε τώρα στην έκθεση που έμεινε από χθε. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση για τον εξορθολογισμό της υλοποίησης του ΔΕΔ του, του, Ευρωπαϊκού, Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ τον κύριο Σέφερ, ο οποίος χρειάστηκε να πάει μια επίσημη στην ε, περιοχή του. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τα TEN. Όπως ξέρετε θέλουμε να υπάρξει απλούστευση των σχετικών project. Ένας κανονισμός ξεπερνά την αρχή της επικουρικότητας στα διάφορα κράτη-μέλη. Εξάλλου, οι περιφέρειες είναι αυτές που δίδουν τις άδειες και προβλέπουν τα συντονιστικά μέσα. Είμαστε λοιπόν να γίνεται ε, σεβασμός των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και να δίδονται οι άδειε ατομικά. Στην ε, συνεδρίαση της ΚΟΤΕΡ είπαμε αυτό για να εξυπηρετούνται καλύτερα και οι πολίτες και αυτό αποφασίσαμε. Σας ευχαριστώ. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο για τη γενική συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν βλέπω να ζητάει κανένας συνάδελφος το λόγο, άρα εξετάζουμε τις τροπολογίες. Έχουμε δύο. Ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία πρώτα απ' όλα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα φτάνουμε στην τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Τελική ψηφοφορία της νομοδότησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε εισηγητά και <coughs> κύριε εκπρόσωπε του εισηγητού. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Τι συνάδελφοι, φτάνουμε τώρα στην τελευταία γνωμοδότηση τη σημερινή συνόδου που παρουσιάζει ο συνάδελφος Φερνάντο Λόπεφ Μύρας για την ψηφιοποίηση στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για γνωμοδότηση πρωτοβουλίας Περιμένουμε τον συνάδελφο. Monsieur le rapporteur, c'est bien Σας δίδω αμέσως το λόγο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μεταξύ των ε, μεγάλων ε, τεχνολογιών εξελίσεων που έχουμε στη σημερινή μας εποχή είναι και αυτό της ε, ε, αύξησης της ηλικίας ζωής. Πρέπει να μπορέσουμε λοιπόν να δούμε νέα πρότυπα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση Αυτές λοιπόν τα νέα αιτήματα μαζί με το έτοιμα ε, όλων μας να έχουμε ισότιμη πρόσβαση για όλους κάνουν απαραίτητο να γίνουν πάρα πολλά στον τομέα της υγείας. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικά συστήματα για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις τις δημογραφικές. Εκτός, από την Εκτός αυτού, η ψηφιακή αλλαγή είναι κάτι που θα βοηθήσει όλους τους επιστήμονες και θα μας βοηθήσει στην πρόληψη ασθενειών την θεραπεία, την διάγνωση και καλύτερη χρησιμοποίηση των δεδομένων στον τομέα της υγείας. Γι' αυτό παρουσιάσαμε την έκθεση αυτή για την ψηφιοποίηση στον τομέα της υγείας και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν με συντονισμένο τρόπο να φέρουν σε πέρα σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής. Το κάνουμε αυτό ζητώντας από όλες τις χώρες και στις περιφέρειες αυτών να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε επιτυχώς το στόχο αυτό. Ο κύριος άξονας, στον οποίο υποστηρίζει, βασίζεται το έγγραφο, είναι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα των δεδομένων όλων των Ευρωπαίων. Για να μπορεί ο καθένας να έχει ε, πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, αλλά να υπάρχουν και οι απαραίτητες ε, υποδομές ώστε να μπορέσουν να ανταλλάσσονται τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια. Γι' αυτό η χρησιμοποίηση ψηφιακών μέσων επιτρέπει την αηφορία και την καλύτερη χρήση των συστημάτων υγείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων και στις προσπάθειες που κατεβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντονίσει τα διάφορα χέλη για την ψηφιακή αλλαγή στον τομέα της υγείας. Είμαστε υπέρ των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων που δημοσιοποιήθηκε χθε. Στο δικό μα έγγραφο όμω προχωρούμε λίγο περισσότερο και προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημιουργία μια πραγματική ιατρικής κλινικής ιστορίας σε ηλεκτρονικό τύπο ώστε να μπορέσουν και ε, διασυνοριακά να ανταλλάσσονται τέτοιου είδου δεδομένα για να μπορέσει να γίνει καλύτερα η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η έρευνα. Και προτείνουμε στον γραφό μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει την δυνατότητα οι γενετικές μελέτες που γίνονται σε ε, ασθενείς να έχουν ένα ε, ειδικό και μοναδικό στοιχείο ε, ατομικό για τον καθένα για να δίδεται συνέχεια σε ό,τι γίνεται. Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή και οι περιφέρειες καλούνται να εργαστούν από κοινού ώστε να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας επιτυχώς την ψηφιοποίηση στον τομέα της υγείας διότι είμαστε πεπιμεσμένοι ότι αυτό είναι κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Και τελειώνοντας θέλω να πω πριν, ε, χωρίς να ξεχάσω να ευχαριστήσω ε, την υποστήριξη που είχαμε στην Επιτροπή μας για να φέρουμε σε πέρα σε αυτήν την εργασία. Η Επιτροπή ΝΑΤ, οι πολιτικές ομάδες, η ε, ομόφωνη συμφωνία που είχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ε, σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και πρέπει να σας πω ότι πιστεύουμε ότι όλες είναι προς βελτίωση του αρχικού κειμένου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ας ανοίξουμε τώρα την γενική συζήτηση όπου έχω ήδη σημειώσει τον κύριο Γιασνάντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Λόπεθ, Πρόεδρο της Περιφέρειας της Μούρθια, για την ε, γνωμοδότηση που αφορά στο παρόν αλλά και στο μέλλον, που αφορά στους προσανατολισμούς ε, του, του ψηφιακού μέλλοντος του συστήματος υγείας προκειμένου να προχωρήσουμε στην καλύτερη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας. Νομίζω ότι η πληροφορία που διαχέεται μέσω των ε, ψηφιακών μέσων μας βοηθούν στην ταχύτητα της ανταλλαγής γνώσης και στο επίπεδο, στο πεδίο της γνώσης θα πρέπει να υπάρχουν και μέσα ελέγχου και εξακρίβωσης της πληροφορίας αυτής αλλά αφορά στους ίδιους τους ασθενείς όπως έλεγε και ο πρόεδρος Λόπεθ Μοίρας. Γιατί εδώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος είναι και ο τελικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών αυτών και όχι το κράτος, όχι κάποιος άλλος τοπικός φορέας. Γιατί με την σημερινή κινητικότητα εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες μπορεί κανείς να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και επομένως πρέπει να μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Επίσης ε, υπάρχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία η τεχνολογία για τα γενετικά στοιχεία που είναι αφορούν και στο μέλλον του τομέα της υγείας. Ήθελα να επιμείνω όμως ότι τα δεδομένα είναι η διοκτησία των ασθενών και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ε, σκοπούς ε, του συστήματος υγείας, του δημόσιου ή του ιδιωτικού στην Βαρακή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερσεν έχει τώρα λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και στην ε, Επιτροπή με μια πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση. Η ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας ε, ε, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας για το μέλλον. Εμείς μπορούμε να, υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε και την γνωμοδότηση και όλες τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί πάντως. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλα μέλη να ζητούν το λόγο για τη γενική συζήτηση και επομένω μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα τις τροπολογίες. Τροπολογία 1 του εισηγητή που αντικαθιστά την αρχική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται δύο τροπολογία υπέρ. Κατά. <coughs> Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. 4 το εισηγητή, αντικαστικά την αρχική 4 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιημένη γνωμοδότηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομοφόνος. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στην ομάδα του. Συνάδελφοι, πλησιάζουμε στο τέλος των εργασιών μας. Μας μένουν ακόμα κάποια λοιπά σημεία. Καταρχάς την εκλογή των μελών του Προεδρείου φαντάζομαι ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις. Εάν δεν έχουμε, θεωρώ ότι έχουμε εγκρίνει. Έχουμε και τα νέα και αναπληρωματικά μέλη. Επίσης προς ενημέρωση στο σημείο. Δεν ξέρω αν κάποιος από σας έχει κάτι για τα διάφορα. Μάλιστα. Να σας πω ότι η επόμενη σύνοδος της Ολομελίας θα είναι εδώ στις Βρυξέλλες, σε αυτήν την αίθουσα, 10 και 11 Απριλίου. Ελπίζω βεβαίως και πιστεύω ότι θα σας δω όλους. 14 και 15 Μαρτίου στο Βουκουρέστι. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή και καλό Σαββατοκύριακο.